Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η πρόεδρός μας, η κυρία Σαρτόρη, ζήτησε από εμένα να αναλάβω την προεδρία σήμερα. Και με αυτή την ιδιότητα σας καλωσορίζω θερμά στην απογευματινή συνεδρίαση γιατί δυστυχώς η πρόεδρός μας η κυρία Σαρτόρη κάπου κόλλησε και θα έρθει καθυστερημένα. Όταν φυσικά έρθει θα της δώσω την Προεδρία και θα την ενημερώσω για τα όσα θα έχουμε συζητήσει μέχρι τότε. Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα με το καθεστώς της διερμηνίας γιατί δεν έχουμε λιθουανικά, σλοβακικά, σλοβενικά και φιλανδικά. Ελπίζω όμως ε, παρά την ε, παράληψη αυτή να καταφέρουμε να διεξαγάγουμε απρόσκοπτο το έργο μας. Ξέρετε, διεξάγονται παράλληλα πολλές ε, συνεδριάσεις και είναι δύσκολο να τις καλύψουμε όλες με πλήρες καθεστώς διερμηνίας. Έχουμε καταρχήν την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας. Η κοινή αυτή συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου, 9 με Το κτίριο Γιάν 4Q2. Αυτά τα διαδικαστικά και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο, το πρώτο σημείο της τη διάταξης, το πρώτο κυρίως θέμα, το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Αντράς Γκιουρκ, απουσιάζει και αντικαθίσταται από τον κύριο Βιντάλ Κουάδρας, στον οποίο και δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εσείς ε, αναπληρώνετε την κυρία Σαρτόρη, εγώ αναπληρώνω τον κύριο Γκιούρκ. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση αντικαταστάσεων και αναπληρώσεων. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, χαίρομαι ιδιαίτερος που μπορώ να αναπληρώσω εδώ τον καλό συνάδελφο και φίλο τον κύριο Γκύρκα και να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το σχέδιο έκθεσής της με θέμα το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζετε τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η χαλιβουργία στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μια και η χαλιβουργία αποτελεί τον πυλώνα των πολλών κλάδων, αυτοκινητοβιγανίας, κατασκευαστικού κλάδου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους αυτούς τους κλάδους. Επίσης απασχολεί 340.000 δημιουργεί 340.000 άμεσες θέσεις απασχόλησης και εκατομμύρια άλλες έμεσες θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου, η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού χαλιβουργικού κράτου... διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην εξασφάλιση της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια στη χαλιβουργία έχουμε χάσει πάνω από 65.000 θέσεις απασχόλησης εξαιτίας απώλειας ανταγωνιστικότητας και ως συνέπεια ε, μιας σειράς παραγόντων. Για παράδειγμα, έχει πέσει ε, αισθητά η ζήτηση του χάλιβα εξαιτία της οικονομικής κρίσης. Δεύτερον, το επιχειρησιακό κόστος ε, της χαλιβουργίας είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με ανταγωνιστές μας από τρίτες χώρες. Και τρίτον, έχουμε λυσαλαίο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, όπως δυστυχώς έχουμε και σε άλλους κλάδους. Γιατί τρίτε χώρες δεν ε, συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα και τι υψηλέ προδιαγραφές και έτσι δεν έχουμε συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού με τους ανταγωνιστέ μα. Εξαιτία λοιπόν της οικονομική και κοινωνική σημασίας ε, της Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο αναχαιτίζοντας την περαιτέρω μετεγκατάσταση του χαλιβουργικού κλάδου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διευρύνοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και βελτιώνοντας τις ε, εργασιακές συνθήκες. Θα πρέπει να τονώσουμε την ζήτηση και να βοηθήσουμε την ε, απρόσκοπτη αναδιάρθρωση του κλάδου. Οπότε το πρώτο τμήμα του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Γκιούρκ επικεντρώνεται σε αυτά τα δύο θέματα. Το σχέδιο έκθεσης ε, τονίζει ότι Επιτροπή και κράτη-μέλη θα θεσπίσουν μέτρα για να τονίσουν τη ζήτηση, να, τηρήσουν τους συναφείς κλάδους, να στηρίξουν τους συναφείς κλάδους και να δημιουργήσουν πρόσφαρες συνθήκες για επενδύσεις. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνεται μια ανάλυση της αγοράς ε, και ένα σύστημα ανάλυση αγοράς το συντομότερο δυνατόν, ώστε να έχουμε διαφάνεια της αγοράς χάλιβα και παλιοσίδερων και να μπορέσουμε να έχουμε σωστούς δείκτες για να μπορέσουμε να εισαγάγουμε τα κατάλληλα μέτρα. Και για να κρατήσουμε ή να προσελκύσουμε ειδικευμένους εργαζόμενους και να αποσοβήσουμε περαιτέρω αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στον κλάδο, θα πρέπει να προβλέψουμε τα κατάλληλα κονδύλια για τη στήριξή του. Αυτό ως προς το πρώτο σκέλος της έκθεσης. Τώρα για το δεύτερο σκέλος της έκθεσης. Ε, επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες ε, και τέσσερις τομείς όπου χρειάζεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Χαέλιβα. Επίσης, ε, για σημαντικές ενεργειοβόρες ε, βιομηχανίες όπως ε, ο Χάλιβας η ενεργειακή τιμή, οι τιμές της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Δυστυχώς είναι πολύ ψηλές οι τιμές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας και μάλιστα το χάσμα αυτό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου το σχέδιο έκθεσης ζητά για άμεση ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, χάλιβα και θα ρίνει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουν μια ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Τώρα, θέμα κλιμα... προστασίας κλίματος και περιβαλλοντικός αντίκτυπο. Είναι μείζωνα σημασία στη συμφιλίωση των κλιματικών και των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον στόχο της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της χαλιβουργίας αποφεύγοντας ε, τον κίνδυνο της ε, διαρροής άνθρακα. Οι διατάξεις ε, για τη διαρροή του άνθρακα θα μείνουν αποτελεσματικές εφόσον κρατήσουμε τη χαλιβουργία στον κατάλογο με τους κλάδους για τη διαφυγή άνθρακα. Αναγνωρίζουμε φυσικά το σημαντικό ρόλο που έχει ο Χάλιβας εξαιτία της αντοχής του και της δυνατότητας ανακύκλωσής του οπότε θα ερήνει την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς παλιοσίδερων και χάλιβα και τη δυνατότητα περισσότερης και καλύτερης ανακύκλωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διεθνείς συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Είναι κέρια σημασία ε, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις να επικρατήσει η αρχή της αμοιβαιότητας ώστε να μην έχουμε ασύμετρες ε, εμπορικέ συμφωνίες, ε, λαθρές αγορές και υπερβολικό έλεγχο ε, τρίτων χωρών για την ροή πρώτων υλών. Και τέταρτο και τελευταίο σημείο, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Αναγνωρίζουμε ότι οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες είναι αναπόδραστες προκειμένου να τηρήσουμε τον στόχο του δικού χάρτη του 2020 για τη μείωση του εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό θα πρέπει να τονώσουμε την καινοτομία με τη χρήση διαρθρωτικών κονδυλίων και να διευρύνουμε τη χρήση νεωτεριστικών μηχανισμών, μηχανισμών καθώς και την αναβάθμιση τεχνολογιών εχμής. Εκ μέρους του κυρίου Γκύρκ του εισηγητή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για την ενεργό συμμετοχή τους στην ε, εκπόνηση της έκθεσης και τις ε, πολύ χρήσιμες ε, παρατηρήσεις τους και τη συνεισφορά τους. Και φυσικά ο εισηγητής περιμένει τις συστάσεις και τις νέες προτάσεις που θα υποβάλλετε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιντάλ Κουάντρας. Σας ευχαριστώ γιατί αναλάβατε να αντικαταστήσατε τον εισηγητή και γιατί μας δώσατε όλες αυτές τις ε, λεπτομέρειες. Οι σκιώδεις εισηγητές δεν είναι παρόντες και αυτοί. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Γαβάς. Επί της ουσίας θεωρώ την ε, πρόταση καλή και σωστή. Η πρόκληση που έχουμε όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στη Χαλιβουργία τονίζεται και πιστεύω πως ε, όλοι μας ε, συμφωνούμε ότι εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τη μεταποιητική βιομηχανία, τη βιομηχανία και τη κατασκευαστική βιομηχανία, χρειάζεται να του δώσουμε προστιθέμενη αξία. Ε, υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Το πρώτο είναι ότι ανάμεσα στα κράτη-μέλη παρατηρείται ανταγωνισμός όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης στη Χαλιβουργία. Ο κ. Σεκάρας ανέφερε τις ε, τιμέ ε, της ενέργειας, επίσης ε, πρέπει να αναφέρουμε τι επιδοτήσεις και πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει μία μείωση της ζήτησης να αυξάνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τις θέσεις αυτές απασχόλησης. Χρειάζεται να βρούμε μία ευρωπαϊκή λύση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να αποφεύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό και να ε, τον αποτρέπουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μεγάλοι όμιλοι στον ε, κλάδο της χαλιβουργίας οι οποίοι βρίσκονται εκτός των συνόρων μας και ηγούνται και θέτουν τους κανόνες. και υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι όμιλοι, οι οποίοι επηρεάζουν κιόλα την βιομηχανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, έπειτα, το θέμα τη αναδιάρθρωση είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. σύμφωνο. Φυσικά και δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε όλε αυτέ τι χαμένε θέσει εργασία στη Χαλιβουργία. Γι' αυτό και χρειάζεται ένα καλό σχέδιο αναδιάρθρωση και την και η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για το σκοπό αυτό. Επίσης πρέπει και τα κράτη-μέλη να ε, δημιουργήσουν και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης ε, της απώλειας θέσεων απασχόλησης. Τρίτο τώρα σημείο και πιστεύω και το πιο σημαντικό είναι η πολιτική καινοτομία. Εξαιτία της ε, παγκόσμιας συγκυρίας για τον ε, Χάλιβα. Παρατηρούμε έναν ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και παρατηρούμε επίσης μια αλλαγή, μια μείωση της ζήτησης ε, λόγω της υπερπροσφοράς και από τη Ρωσία και από την Κίνα και από την Τουρκία και από το Αμπουντάμπι. Και στο Αμπουντάμπι δημιουργήθηκε ένα νέο ε, χαλιβουργείο το οποίο εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιέμαι αν είναι χρήσιμο ή συνετό να εισάγουμε χάλιβα από το Αμπουντάμπι. Όμως έτσι έχουν τα πράγματα και εμείς ε, αυτό που μπορούμε να προτείνουμε είναι η ποιότητα και να προσφέρουμε ποιότητα, ενεργειακή απόδοση και χάλιβα υψηλής ποιότητας. Έχουμε λοιπόν υψηλής ποιότητας χάλιβα, ο οποίος είναι και ε, σταθερός και ευέλικτος και με αυτό το προϊόν στο πλωστάσιό μας ε, μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους υπόλοιπους παραγωγούς. Αυτό λοιπόν πρέπει να τεθεί και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Ήταν το κυριότερο σημείο και τέταρτο ε, σημείο είναι οι εμπορικές σχέσεις. Πρέπει να επανεξετάσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις ε, της Ρωσίας με τον ΕΠΟΕ, ακριβώς λόγω του του ανταγωνισμού, του dumping. Και εδώ πιστεύω πως πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ προσεκτικά πώς ε, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους εταίρους μας στον ΠΟΕ. Ε, δεν γίνεται να καταστρέφονται οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες σε χάλιβα εξαιτίας αυτών των πρακτικών dumping. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουμε πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε αθέμητο ανταγωνισμό, συνεργασία με την Κίνα για παράδειγμα. Ε, ο αθέμητος αυτός ανταγωνισμός δεν λαμβάνει υπόψη του ε, την προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, και μην λαμβάνοντα υπόψη ε, την προστασία του περιβάλλοντο, δημιουργεί λοιπόν αυτέ τι συνθήκε αθέμη του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, όσον αφορά την ε, συμμετοχή των ε, διάφορων αρμοδίων φορέων, όταν ιδρύθηκε η ΕΚΑΧ, υπήρξε μία συμφωνία των ε, τριών ε, μερών των εργοδοτών, ε, των απασχολούμενων και των κρατών μελών που συμμετείχαν. Πρέπει αυτή η συνεργασία να διατηρηθεί και να υπάρχουν ίση όροι και ίση συμμετοχή από όλους. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί πιστεύω, ο τομέας ε, της προστασία των απασχολούμενων και πρέπει να αντλήσουμε από την εμπειρία που είχαμε από την ΕΚΑΧ για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης για τον Χάλιβα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χούσκοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πολύ που συζητούμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή των Μέλλον της Χαλιβουργίας. Διότι πολύ συχνά συζητούμε επιμακρών ζητήματα τα οποία δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την βιομηχανία, με το έργο της Επιτροπής αυτής και χαίρομαι λοιπόν πολύ που τώρα συζητούμε το μέλλον της χαλιβουργίας. Θα ήταν άλλωστε αφελές ε, να μην το κάνουμε. Συζητούμε στα πλαίσια της εκ νέου βιομηχάνησης της Ευρώπης και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλειών. Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό πολύ ικανό στον κλάδο αυτόν. Ο συνάδελφος εισηγητής ανέφερε στο τέλος την ε, καινοτομία ως τελευταίο σημαντικό σημείο στο έγγραφο. Ο Μπέρντ Λάνγκε τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της καινοτομίας και εγώ θα ήθελα να τον στηρίξω. Είναι αποφασιστική σημασία για το μέλλον της χαλιβουργίας η καινοτομία. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφτηκα ένα χαλιβουργείο στη Βόρεια Σουηδία, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. η μονάδα αυτή, να πω ότι είναι ε, μονάδα που παράγει εξαιρετικής ποιότητας χάλιβα, από εξαιρετικής ε, ποιότητας μεταλλεύματα, από ορυχεία που βρίσκονται 300 χιλιόμετρα βόρεια της ε, μονάδας αυτής παραγωγής και η μονάδα αυτή να πω ότι λειτουργεί εξαιρετικά. Η ποιότητα είναι υψηλότερη και είναι μια μονάδα που πραγματικά ξεχωρίζει και βρίσκεται πάνω από όλες τις άλλες μονάδες μαζικής παραγωγής χάλιβα. Αυτές οι μονάδες έχουν συγκεκριμένες ανάγκες εξειδικευμένες ανάγκες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μην ε, συζητούμε γενικότερα το μέλλον, αλλά να επικεντρωθούμε και στις λύσεις σε τέτοιες μονάδες υψηλής ποιότητας. Και αυτό το εργοστάσιο παράγει τόσο υψηλής ποιότητας σε χάλιβα, γιατί, γιατί η καινοτομία είναι υψής της σημασίας, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο αυτό δέχεται παραγγελίες από γερμανικές εταιρείες, από ιταλικές εταιρείες και η μονάδα αυτή διαθέτει επίσης και μία ομάδα προβληματισμού η οποία συζητά συνέχεια νέες μεθόδους ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων χάλιβα. Και επίσης λαμβάνοντας υπόψη και την ενεργειακή απόδοση Δημιουργούν λοιπόν νέα προϊόντα που δεν είναι ζημιογόνα ενεργειακά, είναι χαμηλή σε κατανάλωση. Και να πω ότι είμαι αισιόδοξη για το μέλλον της χαλιβουργίας, με την προϋπόθεση ότι θα αναγνωρίσουμε ότι η χαλιβουργία είναι μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Όπως είπε και ο Μπέρντ Κλάνια, έχουμε εξαιρετικά ικανά άτομα, εξαιρετικά καταρτισμένα άτομα στον ε, κλάδο αυτό, ειδικού εμπειρογνώμονες και αυτοί πρέπει επίσης να προωθηθούν. Αυτό το ταξίδι πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια και μου έδωσε ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη στο μέλλον της Χαλιβουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Σανά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μία έκθεση υπάρχει και δείχνει κάποια πράγματα, κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά σίγουρα δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων, ούτε στο ύψος των σοβαρών περικοπών που θα υποστεί η Ευρωπαϊκή Σιδηρουργία. Αναγράφεται εδώ ε, ο αριθμός των απασχολουμένων, 75.000 είναι μόνο στη Γαλλία. 2% βέβαια των ε, θέσεων απασχόλησης στην βιομηχανία, όμως είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικό το ποσοστό αυτό για την, ε, για τις, για την αυτοκινητοβιομηχανίες, για τις οικοδομές κτλ. Από τις 75.000 το εργαζόμενους, οι μισοί ανήκουν στην εταιρεία Μιτάλ και δεν υπάρχουν όμως εδώ, δεν αναφέρουμε κάποιους μελλοντικού κινδύνους. Λέμε δεν μπορούμε να διατηρήσουμε όλες τις θέσεις απασχόλησης. Γιατί δεν μπορούμε. Εάν έχουμε τα μέσα, θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα πολύ σημαντικά τα οποία τίθενται. Παραδείγματο χάρη, η εξαγορά, η συγχώνευση, η απορρόφηση. Υπάρχει η εταιρεία Μιτάλ, έρχεται αυτός, ο κύριος Μιτάλ, έρχεται στην ε, Ευρώπη, αγοράζει εταιρείε, όχι με τα δεκάτου λεφτά με τις τράπεζες, παίρνει επομένως την επιστήμη, παίρνει την τεχνογνωσία, κλείνει την επιχείρηση μετά και μετά οι χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν το βάρος, το κοινωνικό βάρος αναπολύσεων. Από την άλλη πλευρά, με την αυξημένη ζήτηση από πλευρά της Κίνας, από το 2003 έως το 2010, το 40% του κόστους παραγωγής στο τελικό προϊόν από 40% έχει φτάσει στο 70%. Η παγκόσμια προσφορά και η παγκόσμια ζήτηση αφορά την Κίνα και όταν μειωθεί η ζήτηση από πλευράς της Κίνας και όλες αυτές οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν 100% πρέπει να περιορίσουν την παραγωγή τους, τι θα κάνουν αυτοί. Και στην περίπτωση αυτή η ευρωπαϊκή βιομηχανία, επειδή δεν θα έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, θα κινδυνεύει να πεθάνει. Και αυτό γιατί πριν από την οικονομική κρίση, την πρώτη οικονομική κρίση, η Κίνα είχε 2-3 ε, εκατομμύρια ε, δολάρια σε αποθέματα. Και ενώ πολλές χώρες ε, ε, έχουν φτωχύνει. Τώρα το αποθέματα της ε, Κίνας είναι 4-3 ε, δολάρια και αγοράζει η Κίνα αυτή τη στιγμή όλα τα ανθρακοριχεία και θα αγοράζει και σιδηρουργία. διότι αγοράζει τον άνθρακα, αγοράζει το σίδηρο, έχει φτηνά εργατικά χέρια. Θα μου πείτε τώρα θεμητός ή αθέμητος ανταγωνισμός Αλλά πως να ε, ε, ανταπεξέλθει η Ευρώπη όταν στην βιομηχανία, της, ε, στην δημιουργία δεν υπάρχει κανένα σεβασμός ούτε για το περιβάλλον, ούτε για, τις, για την κοινωνική νομοθεσία και οι ίδιοι οι οι Ευρωπαίοι βιομηχανοί ενισχύουν την μεταφορά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο του γεγονότος ε, της κατάργησης, αν θέλετε, της κοινωνικής προστασίας στον, ε, στην συντηρουργία και πληρώνουμε αυτή τη στιγμή την ενέργεια πολύ ακριβότερα από ό,τι στο παρελθόν. Βέβαια το κόστος ενέργειας δεν είναι το ίδιο παντού γιατί ορισμένες, σε ορισμένες χώρες ήταν δωρεάν η ενεργεία. Ε, η ενέργεια, συγγνώμη. Ε, επομένως θα πρέπει να είμαστε σαφείς, θα πρέπει να λειτουργούμε με ανοιχτά χαρτιά, θα πρέπει να προστατεύσουμε την γαλλική βιομηχανία από επιθέσεις αθέμητες που έρχονται από το εξωτερικό και νομίζω ότι προσπαθούμε να να, εφεύρουμε και να ανακαλύψουμε διάφορα προϊόντα, διάφορες, διάφορα ελάσματα τα οποία ε, είναι καινοτόμα κτλ. Θα τα χάσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ρούμπιχα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία στο μέλλον θα παίξει και θα συνεχίσει να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και όχι μόνο στην Ήπειρό μα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Βιταλ που μίλησε εκ μέρου του εισηγητή κύριου Γκιούρκ. Πιστεύω πω εδώ πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ξανακάνουμε την Ευρώπη ελκυστική για αυτήν την ε, ηγετική βιομηχανία. Η βιομηχανία χάλιβα παίζει πολύ σημαντικό ε, ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και πρέπει λοιπόν να σταθεί στο προσκήνιο των προσπαθειών μας. Ε, τώρα τις προάλλε διάβαζα μάλιστα στην εφημερίδα ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν περήφανος για την ευρωπαϊκή χαλιβουργία και για την μεταφορά χάλιβα και τεχνογνωσία σε προς την Αμερική. Η Χαλιβουργία είναι μια ιδιαίτερα ενεργοβόρος ε, βιομηχανία και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να την συνδέσουμε άμεσα με την ενεργειακή πολιτική, με την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά την ε, μείωση διοξιδίου του άνθρακα, έκκλησης διοξιδίου του άνθρακα από την ε, Χαλιβουργία. Φυσικά Ας μην ξεχνάμε ότι αποφασιστική σημασία έχει εν κατακλείδη ο καταναλωτής, διότι ο καταναλωτής αποφασίζει Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να μπορούν να αγοράσουν προϊόντα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί με χαμηλή παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα και θα είναι όσο το δυνατόν οικονομικότερα. Και ιδιαίτερα τώρα που η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται σε πολύ σημαντική θέση. Ο καταναλωτής θα προτιμήσει να αγοράσει ένα προϊόν που σέβεται το περιβάλλον. Τώρα πιστεύω πως οι υφιστάμενες επιχειρηματικές πρακτικές στον κλάδο πρέπει να σταματήσουν. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις εξαγωγές από την Ευρώπη προς τις τρίτες χώρες και αυτό θα ε, βοηθηθεί μέσω νέων προγραμμάτων έρευνας. Τα προγράμματα αυτά έρευνας θα μας δώσουν τις σωστές βάσεις, τη σωστή προσέγγιση ώστε να γίνει αυτό εφικτό ώστε να δημιουργήσουμε τα καλύτερα και τεχνολογία σε προϊόντα και όχι τα φτηνότερα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας να κάνουμε την αγορά μας και τον κλάδο μας ανταγωνιστικό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον κλάδο και για την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ πολύ καλό που η Επιτροπή Επίτροπος Χέντεγκαρτ ανέλαβε το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, δουλειά του. Πρέπει να τη περισσότερο βέβαια αυτή την έκθεση, γιατί πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την σιδηροβιομηχανία της. Και ε, είναι και θέμα της ιστορίας μας, ιστορικό, το παρελθόν μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ε, συνέπειες ε, όλων αυτών των πραγμάτων. Σαν εισηγητής ε, της οδηγίας ε, για την ε, διάλυση των πλοίων, έδωσα μάχη να, για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα πλοία είναι μία πηγή σιδήρου και χάλιβα που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταλήξει στην Ασία, διότι τα χρειαζόμαστε τα προϊόντα αυτά εμείς. Και διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι το πλοίο η Κώστα Κροτσέρα που είχε προσαράξει στο νησί Τζίλιο θα μεταφερθεί σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι για να διαλυθεί. Και αυτό σημαίνει δεκα, δεκάδες χιλιάδες τόνοι ε, χάλιβα που μπορεί να έχει στη διάθεσή της η βιομηχανία μας. Επομένως υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να ανακυκλώνονται τα προϊόντα διότι με τον τρόπο αυτό χρειάζεται και λιγότερος ε, ανιδρύτης άνθρακα ε, για την παραγωγή και θα ε, στηριχθούμε και όχι τόσο στον άνθρακα αλλά στο υδρογόνο για τις πιο, σημαντικές, πιο σημαντικά στάδια παραγωγής του χάλιβα. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα αυτό, γιατί το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την βιομηχανία και όπως για τον Τάραν, το, το στον Τάραντα στην, στην Ιταλία το έδειξε, πρέπει να είμαστε στην εμπροστοφυλακή, αν θέλετε, των παραγωγών χάλιβα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Πρόντι, είναι συζήτησή μας. Και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο σε έναν εκπρόσωπο της Κομισιόν, εάν είναι κάποιος παρόν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ε, είναι σημαντική ευκαιρία που μου δίνετε να σχολιάσω και να καλωσορίσω αυτή την ε, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Συμμεριζόμαστε πλήρως ε, τις τέσσερις Βασικέ δράσει και του άξονε που προτείνει ο εισηγητή προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Φυσικά, όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, δεν ε, ε, οφείλονται όλα τα προβλήματα στην οικονομική κρίση. Βέβαια, από την κρίση έχουμε χάσει 4.000 θέσεις απασχόλησης, αλλά τα προβλήματα είναι παλιότερα. Ήμασταν οι ε, μεγαλύτερη παραγωγή του χάλιβα. Τώρα έχουμε μόνο το 1% του παγκόσμι, της παγκόσμιας παραγωγής χάλιβα. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στον ανερχόμενο ρόλο της Κίνας που έχει τώρα 50% της παγκόσμιας αγοράς. Επίσης γειτονικές χώρες, Ρωσία, Ουκρανία ή Τουρκία είναι σημαντική ε, παραγωγή. Ε, έχει επανέλθει στο παιχνίδι, έχουν επανέλθει και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επανάσταση σε ό,τι αφορά το σχιστολιθικό αέριο. Θέλουμε λοιπόν ένα ανταγωνιστικό σύστημα ενεργειακών τιμών και μια σωστή συμφιλίωση μεταξύ τη περιβαλλοντική πολιτική και τη επενδυτική πολιτική μα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού και να επενδύσουμε στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Πολύ σημαντική αυτή οι τέσσερι άξονε προτείνει ο εισηγητή και μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής χαλιβουργίας. Να σχολιάσω και δύο ακόμη ε, σημεία που επισήμαναν ε, οι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Σουρούμπεκ ε, υπέβαλε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο για την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πελατών της χαλιβουργίας Βλέπετε ότι στο σχέδιο δράση για τη χαλιβουργία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα μέτρα που προτείνουμε είναι μια προδιαγραφή για το βιώσιμο χάλιβα. Αυτή την προδιαγραφή θα την αναπτύξουμε στο μέλλον και αυτό το πρότυπο, ώστε να μπορέσουν οι πελάτε να κάνουν διάκριση μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων χάλιβα, των κινέζικων προϊόντων και των ευρωπαϊκών, του κινέζικου και του ευρωπαϊκού χάλιβα. Ο κύριο Πρώτη μίλησε για την ανάγκη τη ανακύκλωση των δευτερογενών πρώτων υλών. Ο Horizon 2020 που είναι ε, το νέο πλαίσιο για τις επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη θα ε, χρηματοδοτηθούν πολλές ε, δράσεις, πιλωτικές και προγράμματα που θα έχουν στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης σε πολλούς κλάδους συμπεριλαμβανομένης και της χαλιβουργίας. Εκεί θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για την τόνωση της ανακύκλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση είναι επωφελής για πολλούς λόγους, γιατί και οικονομικά είναι ε, επικερδής και περιβαλλοντικά ωφέλιμη. Γιατί ε, τα πλοία που αναφέρατε που διαλύονται εκτός Ευρώπης πολλές φορές. Αν έχουμε εμείς κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη διάλυση πλοίων θα εξασφαλίσουμε πολύ ποιοτικά υλικά για τους διαφόρους κλάδους της βιομηχανίας μας. Συμφωνούμε λοιπόν με τους τέσσερις άξονες του εισηγητού. Έχουμε κάποια ίσονα σημασία σχόλια, αλλά πραγματικά αφορούν λεπτομέρειες και θα τα διαβιβάσουμε απευθείας στη γραμματεία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βιντάλα Κουάδρας, κύριε αναπληρωτά του εισηγητή, κύριε Γκιούρκα, θέλετε να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπόρεσα να αντικαταστήσω τον κύριο Γκιούρκ στην πρώτη μου παρέμβαση γιατί ουσιαστικά μετέφερε τα δικά του σχόλια. Τώρα, τα σχόλια που θα κάνω τώρα δεσμεύουν μόνο εμένα προσωπικά. Και φυσικά τα σχόλιά μου θα γίνουν με ισπανική προφορά και όχι με ουγγρική προφορά. Κάτι που δεν μπορώ δυστυχώς να αποφύγω. Πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Γκίρκ είναι πολύ καλή. Δεν θα μπορούσε μόνο του να αυτοεπενεθεί, αλλά το λέω εγώ. Γιατί πραγματικά η έκθεση Γκίρκ θέτει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα που επισημάνετε και εσείς συνάδελφοι με τις παρεμβάσεις σας. Σω δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Ναι, μεν έχουμε χάσει χιλιάδες θέσει απασχόληση ε, τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίω. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι από τους σημαντικούς παράγοντες ε, παραγωγής χάλιβα. Μην είμαστε λοιπόν ητοπαθείς και αυτοκαταστροφικοί, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε ισχυρή δύναμη στη χαλιβουργία. Και η ανταγωνιστικότητά μας σε διεθνώς επίπεδο έχει πληγεί ε, σημαντικά. Γι' αυτό έχουμε και χάσει και τόσες πολλές θέσεις απασχόλησης, γιατί οι ανταγωνιστές μας έχουν φτηνότερες τιμές ενέργειας, ε, πολλές φορές ε, εφαρμόζουν αθέμητο ανταγωνισμό στις εμπορικές τους πρακτικές, δεν σέβονται τόσο πολύ, τόσο ευλαβικά όπως εμείς κάποιες κοινωνικές προδιαγραφές, τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, κάποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Έχουμε φυσικά και κάποια εσωτερικά προβλήματα, όπως φοροαποφυγή, αποφυγή, μη πληρωμή ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, οξύτατα, που μας έχουν φέρει στην σημερινή κατάσταση. Πάντως, ο κύριος Γκιούρκ στην έκθεσή του επικεντρώνεται στα σωστά σημεία. Γιατί η ενέργεια αντιπροσωπεύει το 40% του κόστους παραγωγής ε, στη Χαλιβουργία. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια εξασφάλισης ε, πιο προσιτών τιμών ενέργειας. Επίσης, ε, η καινοτομία, η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη είναι νευραλγικές πτυχές του κλάδου. Το είπε ο κύριος και η κυρία Ούσκοκ ότι στην περίοδο αυτή της ε, ε, ιστορικής ε, της ιστορικής περίοδου της Ευρώπης το φως της σοφίας έρχεται από τι χώρε του Βορρά. Μπορεί το φως του ήλιου να επικεντρώνεται στις νότιες χώρες, αλλά το φως της σοφίας εκπορεύεται κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες. Αναφέρθηκε η κυρία Ούσκοκ σε κάποια ατυχή χαρακτηριστικά της Χαλιβοργίας και ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην καινοτομία και στην έρευνα. Πολύ σωστά το είπατε κυρία Ούσκο. Και σίγουρα κατά τη γνώμη μου δεν είναι ο προστατευτισμός η λύση στα προβλήματά μα, Γιατί η εμπειρία μα έχει δείξει πω χώρε που είναι υπερβολικά προστατευτικές ε, βλάπτουν βέβαια κάποιες άλλες, αλλά περισσότερο κακό προκαλούν στον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό και οι εκκλήσεις ε, για περισσότερο προστατευτισμό μπορεί να είναι καλοπροαίρετες, και καλόπιστες, αλλά ε, καλύτερα να αγνοηθούν. Θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και όχι στον προστατευτισμό. Γιατί αν ε, αποδηθούμε σε προστατευτισμό, ουσιαστικά αναγνωρίζουμε την έλλειψη ανταγωνιστικότητάς μας, κάτι που είναι εξαιρετικά επιβλαβές και για την ευρωπαϊκή χαλιβουργία και για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικώ. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι τα σχόλιά μου που ελπίζω θα βρουν σύμφωνο και τον εισηγητή μας τον κύριο Γκιούρκ. Και όπως λέει και ο ίδιος θα πρέπει να συνεχίσουμε και φυσικά και με τη συνεργασία μας, γιατί η Χαλιβουργία είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει και να διορθώσει τα κακό σκήμενα που άνθησαν ιδιαίτερα στην δύσκολη αυτή εποχή της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουιντάλ Κουάντρας. Ισπανο-Ουγγρική συνεργασία για να μπορέσετε να αντικαταστήσετε ε, επάξια τον κύριο Γκιούρκ. Ευχαριστούμε πολύ που μας επιτρέψατε να συζητήσουμε το σημείο αυτό στην ημερησία διάταξη. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών είναι 13 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Δηλαδή, όσον ούπο, δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο για να συντάξετε τις τροπολογίες σας. Τέλος πάντων, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερίας διάταξης, που είναι το σημείο 5, και, ε, δηλαδή εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω την κυρία, Δελκα, κυρία Δελκαστή για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δεύτερη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και τώρα θα συζητήσουμε για δεύτερη φορά την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς μέτρων για την εξασφάλιση ε, κοινού υψηλού επίπεδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα θέμα που συνδέεται άρρηκτα με πολλά από τα θέματα που συζητώνται όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αλλού αυτή τη στιγμή και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον και στην κοινή γνώμη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις 14 Οκτωβρίου, κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψε, επισήμανα ότι στόχος μου είναι να συμβάλλω κι εγώ στην ε, επανεξέταση και αναθεώρηση κάποιων σημείων της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δύο θεμελιώδεις αρχές. Η πρώτη είναι η αρχή της αποτελεσματικότητας και η δεύτερη είναι η αρχή της εμπιστοσύνης. Τώρα, υπό το πρίσμα της ε, πρώτης αρχής της αποτελεσματικότητας, πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε κοινό υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων, ε, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις πτυχές της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής, Επιτροπής Βιομηχανίας, αλλά και της ε, άλλης επιτροπής που έχει υποκλειστικές αρμοδιότητες που είναι η Επιτροπή εσωτερική Αγοράς. Παρ' όλα αυτά όμως ε, έκρινα σκόπιμο να εκφέρουμε και τη δική μας γνώμη στην ε, έκθεση που θα εγκρίνουμε κάποια στιγμή εμείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το δεύτερο παράρτημα προτείνει επέκταση των υποχρεώσεων σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδικτύο, αφήνοντα ανοιχτό το κατάλογο και χωρίς να έχει ακριβείς ορισμούς. Μια τέτοια ανοιχτή πρόταση ενέχει τον κίνδυνο της επιβάρυνσης της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και στη δημιουργία δυσχεριών διαχείρισης εξαιτίας του αριθμού των κοινοποιήσεων ε, συμβάντων, περιστατικών που μπορεί να είναι πολύ υψηλό και πολύ δύσκολο να τον διαχειριστούν οι δημόσιες αρχές σε ένα τέτοιο υψηλό αριθμό συμβάντων εφόσον ε, οι πάροχοι που μπορούν να επέμβουν είναι όλοι οι πάροχοι των δικτύων πληροφοριών. Κατά τη γνώμη μου, έτσι δίνεται έμφαση σε μια διαχείριση που δεν στηρίζεται στον κίνδυνο και άρα δεν ε, επιτρέπει έναν διάλογο και μια αμφίδρομη αξιολόγηση μεταξύ των διαφόρων συντελεστών της αγοράς και των αρμόδιων αρχών. Αν θέλουμε ένα σύστημα πραγματικά αποτελεσματικό, δεν μπορούμε να το στηρίζουμε αποκλειστικά στις κοινοποίησεις. Κατά τη γνώμη μου, οι υποχρεώσεις ε, και οι απαιτήσει που περιλαμβάνονται στο τέταρτο κεφάλαιο θα πρέπει να επικεντρώνονται στις ε, κρίσιμες υπηρεσίες, στις υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών μας, δηλαδή την ενέργεια, τις μεταφορές, την υγεία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Γι' αυτό και υπέβαλα τροπολογία στο παράρτημα 2 και σίγουρα αν υπάρχουν τομείς που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας ε, και οι πάροχοι ε, υπηρεσιών οικειοθελώς ε, θέλουν να κοινοποιήσουν τέτοια περιστατικά συμβάντα, μπορούν να το κάνουν. Αλλά εδώ μιλούμε για υποχρεώσεις. Ποιοι υπάρχοι υποχρεούνται. Περιορίζομαι στις υποδομές ζωτικής σας σημασίας. Στις υποδομές που έχουν κρίσιμη σημασία για τις κοινωνίες μας. Ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες διοικήσεις, το δημόσιο τομέα, είναι σημαντικό να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των δικών τους εφισταμένων υποχρεώσεων, γιατί οι δημόσιες αρχές ασχολούνται με τη δημόσια διοίκηση και το δημόσιο δίκτυο, και φυσικά θέλουμε να δώσουμε μια έμφαση για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Αυτή την ισορροπία προσπάθησα να βρω απαιτώντας από τις ε, κρατικές αρχές να ε, τηρήσουν τις υποχρεώσεις κοινοποιήσεων προβλέποντας το άρθρο 14 αλλά προβάλλοντας ε, τις, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του 15, το άρθρου 15. Κατά τη γνώμη μου, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η Επιτροπή προτείνει την ε, σύσταση μιας αρμόδιας αρχής ε, για την εποπτεία της εφαρμογής της οδηγίας. Κατά τη γνώμη μου, ε, η αποτελεσματικότητα θα προκύψει από την ελαστικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη σε κάθε κράτος υπάρχει ένα ιδιαίτερο μοντέλο στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Σε ορισμένες διοικήσεις έχουμε μια ενιαία αρχή και άλλες, άλλες περιπτώσεις έχουμε τομεακές αρχές. Δεν είναι δόκιμο αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσουμε μια νέα αρχή. Αλλά καλό θα ήταν να έχουμε ένα, νέο, ένα ενιαίο σημείο επαφής ε, που θα είναι ο διάβλος ε, μέσω από τον οποίο θα περνάνε διάφορες πληροφορίες και θα δημιουργείται ένα δίκτυο συνεργασίας, όχι μόνο, όχι είναι αρχή. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο ή την ομάδα αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην πληροφορική, το δίκτυο CERT, και εδώ εφαρμόζω μία παρόμοια λογική. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές υποδομές CERT ομάδων αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ε, πληροφορική. Μερικέ φορέ είναι δημόσιε τέτοιε ομάδε, άλλε φορέ είναι ιδιωτικέ, μερικέ φορέ είναι συνδυασμό των δύο. Έχουν εθνική περιφερειακή εμβέλεια, έχουν ε, κυβερνητική εμβέλεια, καλύπτουν ειδικά τους τομεί και ούτω καθεξής. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει διαφορετικό σύστημα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και εφαρμόζει διαφορετικά κριτήρια τεχνικά και πολιτικά στου ΣΕΡΤ. Ανάλογα με το τι κρίνει σκόπιμο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι ευρωπαϊκέ ομάδε αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην πληροφορική ήδη ε, συμμετέχουν σε διάφορα φόρα και networks, όπω είναι το FACE το Transformation Service. Κατέθεσα τροπολογίες ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η η, τουλάχιστον η παρουσία ενός ΣΕΡΤ ε, για την παροχή οικονομικών ε, ε, παροχή πληροφοριών στους τομείς ζωτικής σημασίας, στους τέσσερις τομείς που σας προανέφερα. Για τους υπόλοιπους τομείς, κάθε κράτος μέλος έχει τη διακριτική ευχέρεια να οργανώνει το σύστημά του όπως το θέλει. Νομίζω ότι η εναρμόνισή μας θα πρέπει να επικεντρώνεται στα απολύτως απαραίτητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την δέουσα ελαστικότητα, ώστε ό,τι λειτουργεί καλά να μην παρεμποδιστεί. Ή να μην εφαρμόσουμε πάση θυσία μία ομοιογενοποίηση αν δεν χρειάζεται. Δεύτερη αρχή, όπως σας είπα, είναι η αρχή της εμπιστοσύνης. Εδώ δεν θα επεκταθώ ιδιαίτερως, γιατί η βασικότερη αρχή κατά τη γνώμη μου, είναι η προηγούμενη αρχή, η αρχή της αποτελεσματικότητας. Τώρα ως προς την αρχή της εμπιστοσύνης έλαβα υπόψη διάφορα θέματα όπως τον αριθμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων που προτείνεται, η συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου στο δίκτυο συνεργασίας, εξαίρεση κάποιων ελέγχων, η εφαρμογή των οδηγιών και στα κοινοτικά θεσμικά όργανα η ανάγκη οι πληροφορίες να είναι αφίδρομες μεταξύ των τομέων που συμμετέχουν και που υποχρεούνται να κάνουν τις κοινοποίησεις και τις ενημέρωσεις ε, που έχουν οι αρμόδιες αρχές. Επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να είναι μονόδρομες ε, αυτές οι πληροφορίες, αλλά να είναι αμφίδρομες. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω, ήδη μίλησα αρκετά. Ελπίζω να απάντησα σε διάφορες απορίες. Περιμένω τις ε, τροπολογίες σας. Τις επόμενες εβδομάδες θα προγραμματίσω και συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις Είμαι πεπισμένη πάντως ότι η συνεισφορά της Επιτροπής μας θα είναι πολύ χρήσιμη, χάρη φυσικά και στη συμμετοχή των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάριν από πλευράς των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου, την κυρία Δελκαστίγιο για την τόσο λεπτομερή έκθεσή της. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια ε, κατεύθυνση και ακολουθούμε την ίδια πορεία συζητώντας ε, αυτήν την έκθεση αυτό που, που, με πειρά, που με κάπως με ενοχλεί ή με κάνει να απορώ είναι αυτή η, ε, η κατανομή ανάμεσα σε επιτροπές του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, ε, καταρχάς ε, συμφωνώ με την προσέγγιση που προτείνει η συγγήτρια. Καταρχάς, όσον αφορά ε, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Προφανώς πιστεύω ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Θα πρέπει να γνωστοποιούν τις, τις διάφορες παραβάσεις. Αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα πρέπει να μιλάμε για τομεί και όχι για υπηρεσίες. Όταν μιλάμε για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα πρέπει ας πούμε, να συμπεριλάβουμε και τις πλατφόρμες πληρωμών ή όχι. Ή όχι. Έχουμε και άλλα θέματα όπως αναφορά το cloud, computing, ε, προσφορά υπηρεσιών. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε ε, μια πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία χωρίς να προχωρήσουμε ε, ε, υπερβολικά. Συμφωνώ εδώ με την ε, κυρία Ντελ Καστίγιο ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση την οποία θα μπορούμε να διαχειριστούμε μετά. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε μέχρι από ποιο βαθμό και μετά ένα περιστατικό θα αναφέρεται. Κάποιες από τις επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν ότι εάν η έκθεση ε, προηγείται του περιστατικού μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο στατιστικά στοιχεία ε, εκ των υστέρων όταν δεν θα υπάρχει το πρόβλημα δηλαδή. Άρα θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση που να επιτρέπει να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση αλλά χωρίς να αυξάνεται η ευαισθησία αν θέλετε και, ε, του συστήματος, να μην γίνεται υπερβολικά ευάλωτο το σύστημα. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα διπλής ροής ενημέρωσης, δηλαδή ε, θα πρέπει να ε, ξέρουμε και το γεγονός αλλά και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει το, η υπεύθυνη υπηρεσία, υπεύθυνος οργανισμός. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάγκη να έχουμε μία ομάδα για να αντιμετωπίσουμε τα κατεπήγοντα 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Και συμφωνώ επίσης με το ενιαίο σημείο επαφής όσον αφορά την αναφορά των περιστατικών Βέβαια, ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε ένα ενιαίο σημείο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν το βλέπω εφικτό ε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον σε κάθε ε, κράτος μέλος να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο. Βέβαια, είναι και θέμα κουλτούρας. Ε, εξαρτάται από την κουλτούρα και, ε, και το σύστημα που εφαρμόζει κάθε κράτος μέλος, γιατί μπορεί να αλλάζει και η προσέγγιση. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια ε, παρόμοια κουλτούρα, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε περιστατικά. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι ίσως να χρειάζεται να συμπεριλάβουμε και κάποια αναφορά στα ανοιχτά διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Sensenelec και την δημιουργία ανοιχτών ελάχιστων προδιαγραφών με κάποιες συστάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Επίσης, να αναφέρω το γεγονός ότι αυτή η οδηγία δεν θα πρέπει να ε, παρακολεί αυτή αυτό, αυτές τις απαιτήσει που έχουμε για την αναφορά προσωπικών δεδομένων στο πακέτο τηλεπικοινωνιών που και εκεί πρέπει να αναφέρουμε περιστατικά. Θα πρέπει να, δημιουργηθεί, ε, να δημιουργηθούν ενιαίες συνθήκες λειτουργίας, αν θέλετε, για όλες τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος και ο ομιλητή, ο κύριος Κρόιτσμαν. Αλλά όμως καταρχάς θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι θα πρέπει να περιοριστείτε όλοι στα τρία λεπτά ως χρόνο ομιλίες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ πρόεδρε. Έχουν υποβληθεί τροπολογίε ε, στι άλλε αρμόδιε επιτροπέ. Ε, γι' αυτό λοιπόν έχει έρθει η ώρα και εμεί να δούμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, με λυπεί ιδιαίτερα η αναφορά στις αποκλειστικέ αρμοδιότητες. Η κυρία Ντελκαστίγιο θα καταρχάς έκανε εξαιρετική δουλειά και γι' αυτό θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Είναι μια πολύ σημαντική βάση για περαιτέρω συζήτηση. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές ε, θέσει ε, στην γνωμοδότηση αυτή. Καταρχά, θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση για το πεδίο εφαρμογή και του ορισμού χρειάζεται μια σύνδεση όλων των ε, φορέων ε, που ε, δρούν στο διαδίκτυο. Επίσης πρέπει να, να επικεντρωθούμε στις λειτουργίες που περιορίζουν και παρεμποδίζουν την επικοινωνία και την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Τώρα, όσον αφορά ε, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον ε, τομέα των μεταφορών, δεν ε, βλέπω τους ίδιους κινδύνους. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων. Χρειάζονται περισσότερες, περισσότερες σημεία επαφής, φυσικά καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι έτσι θα μπορούμε να συνδέσουμε και τα επίσημα και τα ανεπίσημα ε, δίκτυα πληροφοριών, συντονίζοντας τα έτσι κεντρικά. Επίσης, θεωρώ πως είναι σημαντικό στο κείμενο να διατυπώνονται συγκεκριμένοι ορισμοί όσον αφορά τους κινδύνους και τον τρόπο αντιμετώπισης. Η πράξη σε κατεξουσιοδότηση πιστεύω πως ε, είναι κάτι αναγκαίο. Οι προδιαγραφές επίσης χρειάζεται να αναφέρονται σαφώς και πιστεύω πως οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν για μεμονωμένα περιστατικά. Όσον αφορά την αναφορά των περιστατικών, πρέπει και εκεί να υπάρχει κεντρικός συντονισμός. Τώρα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ε, απόρριτο των πληροφοριών στις ε, επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην έχει αυτό συνέπειε συνέπειες στην οικονομία. Χρειάζεται επίσης και πολύ καλή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές όπως είπατε και εσείς, αμφίδρομη πληροφόρηση και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άντερς Ντότερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελ Καστίγιο για την έκθεση και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για την οδηγία αυτή. Το έκανα και στην προηγούμενη συνάντηση έτσι κι αλλιώ. Ε, εγώ αμφισβητώ την ε, διασφάλιση του ε, απορρίτου των προσωπικών δεδομένων. Αυτή τη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίε και κυβερνήσεις ε, στον τομέα της άμυνας χρησιμοποιούν την οδηγία αυτή για τους ε, δικού τους ε, σκοπούς. Ο στρατό είναι επίσης υπεύθυνο. Έχει δημιουργήσει τις κατάλληλε συνθήκες έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί την οδηγία αυτή. Εγώ είμαι υπέρμαχος του Ευρωπαϊκού Project Ειρήνης και σε αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένη η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Πιστεύω πως ε, πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και επίσης να βελτιώσουμε το ζήτημα της διαφάνειας, το οποίο πιστεύω πως ε, αντιμετωπίζεται ελλειπώς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το να δούμε πώς θα παραμείνουν τα δίκτυα ασφαλή. Ε, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις επικοινωνίες και αυτή την εμπιστοσύνη δεν θα την αποκτήσουμε εάν αφήσουμε την ε, φύλαξη και την εποπτεία των δικτύων στα χέρια των κυβερνήσεων, στα χέρια ε, οργανισμών τυποποίησης, τα οποία μπορούν, μπορεί να εγκαθιστούν και κακόβουλο λογισμικό που θα υποκλέπτει τις επικοινωνίες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για τις κυβερνήσεις να, ε, να έχουν αρμοδιότητα ε, στον καθορισμό των ε, προδιαγραφών ασφαλείας. Φυσικό είναι. Επίσης φυσικό είναι να αναφέρεται και η διάσταση της αγοράς και η προστασία των εμπορικών μυστικών. Όμως Πιστεύω πως ε, μια τέτοια κεντρική θέση δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καμία ε, κρατική αρχή. Στη Σουηδία, στη δική μου χώρα, υπάρχει μια εντελώ ανεξάρτητη αρχή Δυστυχώς όμως ο στρατός ε, παρεμβαίνει και επικαλείται την ασφάλεια. Όμως δεν μπορούν να δημιουργηθούν εμπορικές σεζόνες σε εμπόλεμες σεζόνες. Επίσης πρέπει να επανεξετάσουμε το ε, θέμα της διαφάνειας. Η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια εμπιστοσύνης. Ε, δυστυχώς όμως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με αφήνει άφωνη. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω να κατακρίνω την πρόταση αυτή. Πιστεύω πως δεν είναι βασισμένη στην πραγματικότητα και πιστεύω πως πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εμπλεκομένων στην οδηγία αυτή. Βλέπουμε μεγάλη πίεση από όλες τις πλευρές όσον αφορά την ε, ασφάλεια, την στρατιωτική ασφάλεια. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των ειδοποιήσεων, ο μεγάλος αριθμός των ειδοποιήσεων ε, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. ιδιαίτερα, ιδιαίτερα όταν αυτός ο μεγάλος αριθμός ε, αναφορών περιστατικών μπορεί να ε, διακυβεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ε, πολιτών. Και φυσικά οι χειριστές των δεδομένων πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε τα δεδομένα να μην καταλήγουν σε λάθος χέρια, να μην πολλούνται για κέρδος. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ε, τις οποίες ε, διαχειρίζονται όσον αφορά την, ε, τα δεδομένα, οι οποίες ε, δεν διαχειρίζονται με τον σωστό τρόπο και οδηγούν σε ανασφάλεια, τραπεζικές συναλλαγές για παράδειγμα. Όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση του επίπεδου ανασφάλειας, αντίθετο από ό,τι προβλέπει η πρόταση τη Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φόρντ έχει το λόγο. Ο κύριο Φόρντ. Η κυρία Φόρντ. Είσαι ωραίο Ρότζερ, όχι τόσο ωραίο. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τόσο καλή δουλειά που έκανε. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου η ασφάλεια των συστημάτων πληροφόρησης είναι θέμα κλειδί και η Europol μας έδειξε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα, ή μην πω και τρομακτικά παραδείγματα, όπου είχαν ε, τα συστήματά μας, κάποια συστήματα ε, ήταν... Ε, είχε γίνει, είχαν υποστεί hacking και χρησιμοποιηθήκαν με πολύ κακό τρόπο. Θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν τα συστήματα, ε, ποιος τροσόφελος πιανών. Λοιπόν, στο άρθρο 7, ίσως είναι θέμα μετάφρασης, στο αγγλικό κείμενο λέει κάθε τομέας πρέπει να έχει ε, το δικό του σύστημα έρευνας για κάθε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι θέλετε ένα σερτ για κάθε ε, χώρα. δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να αλλάξουμε την διατύπωση. Απ' την άλλη πλευρά, στο θέμα, στο ρόλο της Europol, κατάλαβα ότι επί του παρόντος η επικοινωνία με την Europol γίνεται μέσω της ε, ε, ε, εθνικής αστυνομίας. Δηλαδή η απευθυνόμαστε στις εθνικές αρχές ε, και μετά και εθνικές αρχές απευθύνονται στην ε, Europol. Αυτό θα πρέπει να μείνει φαντάζομαι. Θέλουμε η παρέμβαση της Europol να είναι ευρύτερη, γιατί εκεί μπορεί να έχουμε περιπλοκές. Όσον αφορά τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις, ε, όντως ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία εδώ γιατί τα θέματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα άρα πρέπει να είμαστε σαφείς για το τι αποφάσεις λαμβάνονται και ποιες εκχωρούνται αν θέλετε γιατί δεν θέλω να ε, θέσουμε σε κίνδυνο την διαφάνεια. Τώρα όσον αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στο άρθρο 14. Ξέρω ότι στην ΙΜΚΟ ο εισηγητής πρότεινε να διαγραφεί το δημόσιες αρχές και να μιλάμε μόνο για, τις, ε, ε, για τα market, τους market operators. Ε, εάν θα πρέπει να δούμε ότι αυτοί, αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να είναι υπεύθυνες ανεξάρτητα να ανήκουν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Επίσης, το άρθρο 14 ε, που αναφέρεται το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εξασφαλίσουν να, να ενημερώνονται όλοι. Αυτό το οποίο μπορούν να ξέρουν ή να κάνουν μάλλον είναι ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί έτσι ώστε να υπάρχει η ενημέρωση. Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ενημέρωση αυτή καθεαυτή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Και εδώ θα ήθελα να διευκρινιστεί κάπως η διατύπωση. Για το άρθρο 16 υπάρχει μία ανησυχία από πλευράς του κλάδου για τα πρότυπα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα αναφορών ή όχι. Συμφωνούμε με την διατύπωση, ίσως ότι θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά αυτό το οποίο θέλουμε δηλαδή να γίνεται στην Ευρώπη θα πρέπει να το συνδέσουμε με αυτά τα οποία γίνονται και, στους, και στα άλλα σημεία του πλανήτη. Τέλο πάντων, αυτά νομίζω καταρχά. Υπάρχουν κάποιε μικρέ μικρές διορθώσει, ε, αλλά θα νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι τώρα. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπή, το είχα πει ήδη και στις 14 Δεκάτου, όμως πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει σε συμβιβασμούς που καθιστούν την πρόταση αποσπασματική και εν τέλει αναποτελεσματική. Φοβούμε ότι η τελική πρόταση περισσότερο εξυπηρετεί τις ανάγκες της γραφειοκρατίας της Επιτροπής δηλαδή το να περιφρονήσει ο κάθε επίτροπος από ένα πεδίο δραστηριοτήτων, cyber security, cyber crime, cyber war, παρά το να δημιουργήσει μια συνολική ευρωπαϊκή λύση που θα διασφαλίζει τα ασφαλή πληροφοριακά δίκτυα που οι κοινωνίες μας και οι οικονομίες μας έχουν ανάγκη. Μόλις τον τελευταίο μήνα είχαμε δύο μεγάλες κλίμακας επιθέσεις σε στόχους που θα περίμενε κανείς ότι γνωρίζουν καλά να προστατεύουν τους εαυτούς τους, των οποίο είναι σαφές ότι το μέγεθος και οι επιπτώσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένες εθνικές υποθέσεις. Στην επίθεση της Vodafone στη Γερμανία είχαμε απώλεια στοιχείων για δύο εκατομμύρια Γερμανούς πολίτες. Στην επίθεση στην Αμερικανική εταιρεία Adobe χάθηκαν τα στοιχεία 38 εκατομμυρίων πελατών, μεταξύ των οποίων και πολλών Ευρωπαίων, και όχι 2,9 όπως οι ίδιοι ψευδώς είχαν ανακοινώσει πριν λίγες μέρες. Και κυρίως οι hackers απέκτησαν πρόσβαση στον πρωτότυπο προγραμματιστικό κώδικα που θα τους επιτρέψει στους επόμενους μήνες να πραγματοποιήσουν πολύ πιο στοχευμένες και μαζικές επιθέσεις. Φοβούμε ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι λύσεις που επιλέγει η Επιτροπή μπορούν να εξυπηρετούν την ίδια την Επιτροπή και να καλύπτουν τα ισχυρότερα κράτη-μέλη που έχουν ή νομίζουν ότι έχουν τους δικούς τους ισχυρότερους μηχανισμούς προστασίας του διαδικτύου. Ωστόσο, όπως μπορεί να σας πει ο κάθε ειδικό, η ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος είναι όση ακριβώς είναι η ασφάλεια του πιο αδύναμου κρίκου του. Όποιος στην Ευρώπη νομίζει ότι τα δικά του δίκτυα είναι θωρακισμένα και ότι δεν χρειάζεται ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και συντονισμός, κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη όπως και με την οικονομία. Κλείνοντας να αναφέρω ότι εξακολουθούμε να δημιουργούμε αυτόνομες ad hoc δομές, όπως είναι το EU CERT, την ίδια στιγμή που ο ΕΝΙΖΑ θα μπορούσε να αναλάβει ακόμη σημαντικότερο συντονιστικό ρόλο και κυρίως να βοηθήσει τα μικρότερα κράτη-μέλη να θωρακίσουν τις δικές τους κρίσιμες υποδομές. Ήδη η κυρία Ντελκαστίγιο έχει καταθέσει με το report της μερικές ουσιαστικές βελτιώσεις. Στην ίδια κατεύθυνση και με όσα προανέφερα θα κινηθούν και οι δικές μου τροπολογίες και εύχομαι να μην δούμε ξαφνικά να αναδύεται στην επιφανειακή οικονομία το deep internet, τα λογισμικά τώρα ή τα bitcoins. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Thank you. Next time. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έλμερ. Uh, well, thank you, uh, Mr. Chairman. and all. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω φυσικά στην εισηγήτρια, αλλά πρώτα να κάνω μια σκέψη και ένα σχόλιο μετά την ε, μακροσκελή εκτενή ε, παρέμβαση κυρία Σαντερστότερ. Όπως λέμε στην Αγγλία, όχι θα την γλιτώσει κανείς επειδή είναι παρανοϊκός, ε, οπότε νομίζω να αξιοποιήσουμε αυτές τις πολύ χρήσιμες συμβουλές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγητή για το έργο της, για την γνωμοδότησή της και να επισημάνω το σχόλιο της ότι προτιμά τη συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών αρχών, αν κατάλαβα καλά, παρά τη δημιουργία μιας νέας ε, πανευρωπαϊκής αρχής. Εμείς ε, ε, είχαμε τον Τζον Major, όταν είχαμε τον John Major πρωθυπουργό και είχε πει κάτι παρεφερές με αυτό που θα πω εγώ. Όταν η απάντηση είναι περισσότερη γραφειοκρατία, τότε η ερώτηση που έχουμε θέσει είναι σφαλμένη. Θεωρώ σαφές ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών και το, η δικτύωση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι ε, αποτελεσματική, στενή και σίγουρα είναι και λιγότερο δαπανηρή από τη δημιουργία μιας νέας γραφειοκρατικής δομής. Γι' αυτό συμφωνώ με την σχετική πρόταση συγκήτριας για την καλύτερη συνεργασία των κρατικών αρχών και όχι τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δομής. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Τζουζέπε Μπεμόντε και είμαι τη μετάρχης ε, ε, της, ε, της Μονάδας για την Ασφάλεια των Δικτύων στην Αρμόδια Γενική Διεύθυνση και ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις πολύ καλές προθέσεις της και το σκεπτικό της γνωμοδότησής της. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Η έκθεση περιλαμβάνει και κάποιες ιδέες που θα μας βοηθήσουν κατά πάσα πιθανότητα να επιλύσουμε κάποια δύσκολα προβλήματα, ή κάποια εμπόδια που έχουμε και στο Συμβούλιο. Για παράδειγμα, δεν είμαστε κατά της πρότασης για περισσότερες, ε, περισσότερα σέρτη, περισσότερες εθνικές αρχές. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε ένα ενιαίο σημείο επαφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πιστεύουμε ότι οι προτάσεις έκθεσης για, το ε, το, για τη φύση της πληροφορίας ε, που δεν θα πρέπει να είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες που κυκλοφορούν στα δίκτυα είναι πολύ λογική ιδέα. Επίσης, οι προτινόμενοι κανόνες για τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση των ε, διαφόρων περιστατικών παραβίασης θα πρέπει να εξεταστούν πολύ φυσικά πιο ε, εδελεχώς, αλλά εκ πρώτης όψης φαίνονται λογικά τα σχόλια της ε, εισηγήτρια και προτάσει. Ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Έλμαρ, νομίζω ότι έγινε μια παρεξήγηση εδώ. Εμείς δεν προτείνουμε τη σύσταση μιας νέας αρχής, προτείνουμε ένα μηχανισμό συνεργασία. Όταν ε, εκπονήσαμε την μελέτη επιπτώσεων, αποκλείσαμε την ιδέα τη σύσταση μια νέα αρχή που θα είναι αρμόδια για την ασφάλεια των δικτύων στην Ευρώπη. Απλώ θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό συνεργασία που θα συνδυάζει τις υπάρχουσες δομές ασφάλειας των δικτύων και τις νέες, γιατί δεν έχουν όλα τα, χαρ... κρατη μια τέτοια δομή αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των δικτύων και ε, βελτιώνουμε την συνεργασία μεταξύ τους με το μηχανισμό που Τώρα, εκεί που διαφωνούμε με την εισηγήτρια είναι η εμβέλεια της διαχείρισης ε, του κινδύνου και της υποχρέωσης ε, κοινοποίησης των διαφόρων ε, συμβάντων ασφαλείας περιστατικών. Η εισηγήτρια προτείνει περιορισμό του πεδίου εφαρμογή και περιορισμό των υποχρεώσεων αποκλείοντας αυτούς τους internet neighbors που λέμε. Έχουμε όμως κάποιες ε, εταιρείες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ατζέντα και κατά τη γνώμη μου θα ήταν σφάλμα να τους αποκλείσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, για παράδειγμα, οι εταιρείε αυτές πραγματικά διαδραματίζουν ένα ζωτικό ρόλο στο ψηφιακό θεματολόγιο. Γιατί παρέχουν υπηρεσίες ε, επικοινωνίας και πληροφορικής, οπότε έχουν άμεσο ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές ε, τηλεπικοινωνίες και επίσης ε, δημιουργούν μια πλατφόρμα που είναι πολύ σημαντική, όπως οι μηχανές αναζήτησης ή οι πλατφόρμες κατανομής περιεχομένου, που είναι πολύ σημαντικές στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε. Οπότε οι εταιρείε αυτές βρίσκονται στην καρδιά του ηλεκτρονικού εμπορίου ουσιαστικά και επίσης παρέχουν πόρους ε, που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια και τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτύου. Κάτι που ε, αναφέρθηκε είναι η ανάγκη των ε, συνθήκων ισότιμου ανταγωνισμού. Με βάση το άρθρο 13α της Οδηγίας Πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, παραδοσιακή πάροχή πάροχη υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και δικτύων υπόκεινται στις υποχρεώσεις ε, δικτύου και πληροφορίε, δηλαδή διαχείρισης του κινδύνου και κοινοποίησης ε, των περιστατικών. Μερικές από τις ε, εταιρείες όμως μπαίνουν σε αγορές που κατά παράδοση περιορίζονται σε βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών. Επίσης δεν έχουν έδρα σε ε, χώρα. Είναι κυρίως αμερικανικές εταιρείες. Θα ήταν λάθος και κρίμα να τις αποκλείσουμε ε, και από την υποχρέωση διαχείρισης κινδύνου και κοινοποίηση περιστατικών. Γιατί έτσι δεν θα ε, εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε πραγματικά ισότιμο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να έχουμε μια οδηγία που θα αντέξει και στο μέλλον. Γιατί αν ε, αποκλείσουμε αυτές τις εταιρείες και περιορίσουμε τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και διαχείριση του κινδύνου σε ορισμένου πολύ σύντομα η οδηγία θα ξεπεραστεί από, τα, από, τις, ε, από το μεταβαλλόμενο κόσμο και θα γίνει ουσιαστικά παροχημένη και παρχιομένη πριν καν τεθεί σε ισχύ. Ευχαριστώ. Η συγκεκριά μα τώρα, κυρία Πιλάρ Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, επειδή αφιερώσαμε ήδη μεγάλο τμήμα της απογευματινής συνεδρίασης ε, στη δική μου γνωμοδότηση, θα περιοριστώ στη δευτερολογία μου σε λίγες μόνο παρατηρήσεις. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές που έλαβαν το λόγο για την προθυμία που έδειξαν και το συνεργάσιμο πνεύμα τους. Ε, όλες σχεδόν ε, οι παρεμβάσεις ε, έδειξαν ότι υπάρχει περιθώριο για σύγκληση. Θα το δούμε και στην εξέταση των τροπολογιών, αλλά πιστεύω ότι γενικά ο προσανατολισμός μας είναι κοινός. Η κατεύθυνσή μας είναι η ίδια. Οπότε έχω προέστημα καλό και πιστεύω ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, στην πρόταση οδηγίας ε, θα είναι πολύ θετική και θα βοηθήσει πολύ στην διαμόρφωση της οδηγίας. Δεν θα αναφερθώ λεπτομεριακά στις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Μερικές φορές ε, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πιστεύω ότι θα τις λύσουμε και θα καταφέρουμε να βρούμε μία κοινή γραμμή. Ακόμη και δεν υπάρχει απόλυτη σύγκληση, τουλάχιστον ε, να συμφωνήσουμε ως προς την κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστροπή για την πρότασή της, γιατί ανέλαβε τεράστιες ευθύνες ε, και ε, οι προκλήσεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι τεράστιες, γιατί οι προκλήση στον τομέα της ενέργειας, της υγείας ή σε άλλους τομείς που δεν αναφέρονται στα δίκτυα είναι παλιά θέματα, δεν είναι καινούργια, οπότε οι προκλήσεις είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Τώρα, εδώ, στα ψηφιακά θέματα, μπαίνουμε σε παρθένο έδαφο, ουσιαστικά. Και οι προτάσεις ε, είναι πολύ πιο εξεζητημένες, οι προκλήσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την πρότασή της σε πραγματικά καινοτόμα ζητήματα και νεοτεριστικά. Σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε ότι δεν προτείνεται τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Αρχής. Ναι, μεν, αλλά προτείνεται μία ενιαία αρχή σε κάθε χώρα μέλος. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι ακριβώς εξαιτίας της ποικιλομορφία της οργάνωσης ε, των μηχανισμών ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στα κράτη-μέλη, καλό θα ήταν να σεβαστούμε τις παραδόσεις αυτές και τις οργανώσεις που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη και να εφαρμόσουμε κάποια ελαστικότητα. Να έχουμε ενιαία σημεία επαφή ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά όχι μία και μόνο αρχή σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, Κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και βρίσκεται στην καρδιά της συζήτηση είναι το εξής. Ποιος συμμετέχει σε όλα αυτά, ποιος φέρει την ευθύνη ώστε να πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογή. Ποιοι κλάδοι. Οι εταιρείε του διαδικτύου, οι επιχειρήσει του διαδικτύου, ποιε άλλε επιχειρήσει. Επιχειρήσει λογισμικού, software, hardware, γιατί δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση Ευρωπαϊκής επιτροπή; Ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν αυτές τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και διαχείριση κινδύνου. Επίσης, οι ευθύνε τους ε, στη λειτουργία των δικτύων. Ποιες είναι, γιατί αν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνε τους, δημιουργούν προβλήματα και στους παρόχους ε, υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Ποιους θα περιλάβουμε λοιπόν και ποιους θα αποκλείσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα και θέλοντας να εξασφαλίσουμε ε, την μέγιστη ασφάλεια του δικτύου, μερικές φορές αντί να επικεντρωνόμαστε στα ουσιώδη, προτιμούμε να καλύψουμε όσο το δυνατό περισσότερους. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Και ποια είναι τα ουσιώδη, είναι οι υποδομές ζωτικής σημασίας. Αυτό θα ήταν ήδη ένα τεράστιο βήμα και ο χρόνος θα δείξει ε, αν είναι δόκιμη αυτή η οδηγία, γιατί σίγουρα δεν θα εξαντλήσει η οδηγία αυτή όλο το θέμα της ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών. Απλώς, ε, αν επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους τομείς, θα συνδυάσουμε την αποτελεσματικότητα με την εμπιστοσύνη. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Επίσης, θα εφαρμόσουμε μια ελαστικότητα και θα σεβαστούμε τις οργανωτικές δομές των κρατών μελών για τα θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Με όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα κάνουμε ήδη ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Δεν θα είναι το οριστικό βήμα, το τελικό βήμα, αλλά θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και αυτή τη στιγμή αυτό ζητά από εμά η κατάσταση. Ένα περιορισμό του πεδίου εφαρμογής, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη. Και φάνηκε από τη συζήτηση ότι περισσότεροι συνάδελφοι προ αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μα και είμαι βέβαιη ότι θα βελτιώσουμε σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις, ε, ε, τις παρατηρήσεις και για τα καταληκτικά σας σχόλια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 12 Νοεμβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμή για την υποβολή των τροπολογιών. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι τα μέτρα για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας. Καταρχάς θα δώσω τον λόγο στην κυρία Edith Χερτσκοντ, την εισηγήτρια. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε και τη δική μου έκθεση για την αποτελεσματική χρήση των ε, υποδομών και την ανάπτυξη λύσεων. Χρειάζεται η λύση που θα βρεθεί να επιταχύνει και να διευκολύνει την, ε, τις ψηφιακές υποδομές για όλους. Και πώς θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να βρούμε συνέργειες και συνεργασίες και να απομακρύνουμε τα εμπόδια. Κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η πρόταση της Επιτροπής είναι η αύξηση της συνεργασίας μέσω γραφειοκρατίας, διευκολύνοντας την διαδικασία διοδότησης, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές. Και αυτό δεν είναι ξαφνικό. Αν δείτε τι έγινε με το ε, Λονδίνο ή με την υπόθεση απο, ε, αποχέτευσης της Βαρκελόνης, θα δείτε ότι υπάρχει κάποιο προηγούμενο, όπως επίσης και σε άλλες χώρες, τη Γερμανία, τη Δανία και τη χώρα μου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαλέγει τα καλύτερα παραδείγματα από τις διάφορες χώρες και τα παρουσιάζει ταυτόχρονα και μαζί. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μία λύση γρήγορη, διότι δεν μπορούμε διαφορετικά να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα όσοι ζουν στην Ήπεθρο, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους παρέχουμε αυτές τις ψηφιακές υποδομές. Και ε, έχοντας ακούσει και την προηγούμενη συζήτηση, πρέπει να πω ότι οι κάτοικοι της Ήπεθρου έχουν και εκείνοι το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμπεριληφθούν στις ε, συζητήσει ε, αυτέ ε, για την ψηφιακή ασφάλεια. Φυσικά δεν μπορείς να έχεις ψηφιακή ασφάλεια αν δεν έχεις και πρόσβαση. Και χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί αυτή η πρόσβαση. Η Ευρώπη θα γίνει περισσότερο ανταγωνιστική μόνο με την διόρθωση του προβλήματος αυτού, της πρόσβασης. Στα πλαίσια του, δημοσιονομ... του σε δημοσιονομικού πλαισίου δεν διατίθενται ε, κονδύλια για αυτό το σκοπό. Έχουμε λοιπόν περιορισμένες ε, νομικές ε, δυνατότητε για εύρεση λύσης. Με χαρά μου λοιπόν είδα ορισμένε από τι τροπολογίε που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Με μεγάλη μου έκπληξη τις είδα αυτές τις τροπολογίες και επίσης αξεπλάγει με το πόσο συχνά συνάδελφοι από πολύ διαφορετικές πολιτικές ομάδες με πολύ διαφορετικές απόψεις υπέβαλαν παρόμοιες τροπολογίες. μια πολύ, ε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός τροπολογιών ζητά κανονισμό αντί για οδηγία. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί η οδηγία θα ήταν μια πιο γρήγορη λύση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Απορώ με όσους κατέθεσαν αυτή την τροπολογία διότι ένας κανονισμός μας δίνει μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ελαστικότητα και μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής. Και είναι και υποχρεωτικός ούτως ή άλλως, οπότε δεν μπορούν να αποφύγουν την εφαρμογή του. Απορώ λοιπόν με τους συναδέλφους που θεωρούν ότι η οδηγία είναι καλύτερη και γρηγορότερη λύση από έναν κανονισμό. Συμφωνώ με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι χρειάζεται καλύτερα κανονισμός και γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για τις συμβαστικές τροπολογίες θα προσπαθήσω και θα συνεχίσω να, προσπαθήσω, να προσπαθώ να βρεθεί λύση. Υπάρχουν ε, πολλές τροπολογίες για εξαιρέσει για το ποιες υποδομές θα πρέπει να εξαιρούνται και γιατί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα πραγματικά να με βοηθήσετε να καταλάβω γιατί αναφέρονται αυτές οι μερικές εξαιρέσεις. Γνωρίζω ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι βέλτιστες πρακτικές δείχνουν ότι, ένα, ότι οι συνέργειες δημιουργούνται με τη συνεργασία. Και θα ήθελα επίσης να, την προσοχή, να επιστήσω την προσοχή σας στις τροπολογίες που αφορούν την ασφάλεια. Ιδιαίτερα για τον τομέα αυτό καλωσορίζω όλες τις τροπολογίες που ζητούν περισσότερη ασφάλεια. Αντίθετα με τις τροπολογίες οι οποίες ζητούν μεν ασφάλεια, δεν θέλουν όμως να τροποποιηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός σε αυτών τον δύο ειδών τροπολογίες. Η πρόταση λοιπόν για συνέργειες και αυξημένη συνεργασία, αυτές ε, με βρίσκουν σύμφωνοι, αλλά οι τροπολογίες ε, της άλλης κατηγορίας με βρίσκουν τελείως ε, αντίθετη και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λοιπόν. Επίσης πιστεύω πως είναι σημαντικό να αναφερθούμε στον ορισμό της υψηλής ταχύτητας αυτό ήταν και ένα από τα δυσκολότερα ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσουμε. Να σας πω ότι δεν αρκεί μόνο να δώσουμε έναν ορισμό για την υψηλή ταχύτητα. Γιατί οι ταχύτητες μεταβάλλονται με την πρόοδο της τεχνολογίας. Κάτι που θεωρείται υψηλή ταχύτητα σήμερα μπορεί να είναι πολύ αργό αύριο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσαρμοζόμαστε και στα επόμενα χρόνια να φροντίσουμε να περάσουμε από τις παθητικές υποδομές στις ενεργητικές υποδομές. Σίγουρα πρέπει να κυμαίνονται από τα 50-100 αλλά όπως είπε και ένα συνάδελφος, η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συζητήσουμε το θέμα του ορίου των 100 Mbit σήμερα έτσι ώστε όταν θα αναθεωρηθεί ο οργανισμός, ο κανονισμός, συγγνώμη, να μπορούμε να τον προσαρμόσουμε με αναθεώρηση. Να μπορούμε να περάσουμε εύκολα δηλαδή από μια ταχύτητα 100 Mbit σε μια ταχύτητα 1 Gbit. Ίσως είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο και σίγουρα δεν θα διαφωνούσαμε κάποιον που θα ζητούσε αύξηση του όριου ταχύτητας αλλά η λύση που έχω να προτείνω είναι αυτή. Επίσης, συζητήσαμε εκτενώς τις ε, συνθήκες για συνεργασία. Δεν πιστεύω όμως ότι ο κανονισμός αυτός στοχεύει στην αντικατάσταση των διαπραγματεύσεων για τους ε, πλεκομενούς φορείς. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα είτε να βρουν μια λύση είτε να αρνηθούν την συνεργασία εάν οι ε, όροι δεν είναι ευνοϊκοί. Αλλά αυτό πιστεύω πως ε, δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς και δεν θα έπρεπε να το λύσουμε εμείς. Αυτή είναι εδώ την ε, πρόταση. Είναι όμως κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και να το συζητήσουμε αργότερα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη μου χαρά είδα ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, έστειλε μια επιστολή στο Συμβούλιο και με χαροποίησε πολύ το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Συμβουλίου το οποίο Συμβούλιο δεσμεύτηκε για την ψηφιακή εσωτερική αγορά και την ε, επέκταση των ψηφιακών υποδομών. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα ότι μέσα σε αυτή την νομοθετική περίοδο θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και γι' αυτό λοιπόν ελπίζω εγώ και οι υπόλοιποι σκιώδεις συζητητές να βρούμε μια ε, λύση για όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση ο κύριος Χόκμαρ είναι ο πρώτος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω εκεί, σαν τα παλιά. Πολλά έχουν βέβαια συμβεί έκτοτε. Ευχαριστώ και την κυρία Χέρψοκ για την παρουσίασή της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι όταν μιλάμε για όλο αυτό το project, ο στόχος είναι να αυξήσουμε το δυναμικό και τις ευκαιρίες. Και ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτά τα πλαίσια να συμφωνήσουμε και πάνω στο γεγονός ότι το 2020 και η ε, οι συν, γρήγορες δεν θα είναι 30 ή 100 Mbit, τα, ε, ίσως Αυτά είναι προκλήσεις ε, του σήμερα και όχι του αύριο και ο βασικός στόχος όλων αυτών των συζητήσεων είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σε ηγετική θέση. Άρα θα πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά τις ανάγκες για υψηλές ταχύτητες και η, ανα... Ε, ε, οι αλλαγές ε, τις οποίες ανέφερε η κυρία Χέρτσοκ είναι ουσιαστικές, είναι απαραίτητες, γι' αυτό θα πρέπει να αφήσουμε τους παλιούς στόχους πίσω. Και αυτό το λέω, διότι όταν μιλάμε για ευρυζωνικά συστήματα, όσο και αν ουδέτεροι πρέπει να είμαστε όσον αφορά την τεχνολογία, θα στηριχθούμε σε, μία, σε ένα συνδυασμό ο, σταθερής και κινητής μεταφοράς ευρυζωνικής ε, ε, επικοινωνίας. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα γιατί και για τις ίνες, οπτικές ίνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της συζήτησης ε, και της πρότασης. Η πρόταση αυτή κανονισμού την χάνει σοβαρής υποστήριξης από τα μέλη της ε, Επιτροπής που θέλουν να γίνει μια οδηγία. Και γι' αυτό γιατί. Γιατί η ανάπτυξη της ε, βριζονικής επικοινωνίας δεν είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι στόχο των κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε πώ οι εταιρείε, οι κοινότητε, όλοι αυτοί Τέλο πάντων θέλουν να, να το προωθήσουν. Κάποιε κάποιες φορές είτε ανταγωνιστικά είτε μέσα στα πλαίσια μιας συνεργασίας. Αλλά εκεί ανήκει η αρμοδιότητα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Άρα ο στόχος μας δεν είναι να μπούμε σε λεπτομέρειες και να ρυθμίσουμε σε λεπτομέρειες το όλο σύστημα. Διότι το κάθε περιβάλλον, κάθε κρότη χώρα είναι διαφορετική και από γεωγραφικής πλευράς, από το κλιματικής πλευράς, από την απόσταση και κυρίως όσον αφορά την νομοθεσία αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η νομοθεσία. Υπάρχουν διαφορές για το πώς ε, προωθείται η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων σήμερα και πιστεύω ότι είναι, υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της οδηγίας, υπέρ της ύπαρξης μιας οδηγίας. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι έχουμε τους στόχους, οι στόχοι πρέπει να είναι οι ίδιοι, αλλά θα επιτευχθούν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος μέλους. Και κάνοντας κάτι τέτοιο, διασφαλίζουμε ότι τα κράτη-μέλη καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε τα πράγματα να είναι εύκολα, όσο να τον πιο εύκολα για τις εταιρείε, για τους δήμους της κοινότητας και για τους διάφορες, διάφορους παράγοντες, να συνδυάσουν και να χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες δομές, χωρίς να μπλέκονται σε άλλα χωράφια νομοθετικά. Ε, ε, υπάρχει το σύστημα διανομής νερού, ας πούμε, παραδείγματος οι νομικές ε, δομές τις οποίες θα πρέπει να σεβαστούμε, δηλαδή θα πρέπει να αντλήσουμε παραδείγματα και από άλλους τομείς. Και θα πρέπει αυτό να γίνει όσο δυνατόν, με όσο δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία και με πιο σαφείς στόχους. Ένα παράδειγμα που νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε από, άλλες, από άλλη προοπτική. Ας πούμε, εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές ε, ε, ε, με επισήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε, να λέμε ότι αυτό είναι υψηλό σύστημα, υψηλής ταχύτητα σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε αυτό είναι ένα σπίτι αν θέλετε ή ένα κτίριο υψηλή ταχύτητα. Ε, είναι σαν να λέμε ας πούμε αυτό είναι ένα, σύστημα, ένα σπίτι όπου έχει ηλεκτρικό. Είναι ξεπερασμένο, δηλαδή θα είναι ξεπερασμένο κάποια στιγμή αυτό. Άρα είναι σημαντικό να ε, υιοθετήσουμε και να εξασφαλίσουμε ένα στοιχείο το οποίο αναφέρει το κείμενο της Κομισιόν που είναι η διασφάλιση ε, σωστού ανταγωνισμού ανάμεσα στις, ε, στους διάφορους εμπλεκόμενους. Και, για την έκθεση, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται συχνά και στην έκθεση κυρία Χέρτζο και τις, τις τροπολογίες. Γι' αυτό, Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητάμε το κείμενο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι μια οδηγία και να δεν θα πρέπει να είμαστε ε, να μπούμε σε πολλές, πολλές λεπτομέρειες ε, και να είμαστε κατευθυντικοί αν θέλετε, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά τους στόχους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κολακία νομίζω ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Κύριε αν θέλετε το λόγο.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 το θέμα είναι να έχουμε ένα ευρύτερο ανταγωνισμό για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλο το δυναμικό του κλάδου. Ποια είναι η γνώμη της ηγήτριας ε, για τις επιμέρους ε, συμβαστικές προτάσεις. Θεωρεί και η συγγήτρια ότι το δίκτυο θα πρέπει να είναι όσο πιο ανοιχτό γίνεται και να περιλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες. Αυτό είναι και προς όφελος των χρηστών. Ευχαριστώ κυρία Δότερ. Ευχαριστώ. Και... Ε, εξετάσαμε τις τροπολογίες και χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία και κοινοί παρανομαστές. Δεν είναι σωστή πρόταση κανονισμού, γιατί είναι το πιο δεσμευτικό νομοθετικό όργανο της κοινότητας για την ε, λεπτομεριακή ρύθμιση και των τοπικών ε, προβλημάτων και αρχών. Βέβαια, άκουσα ότι οι υπάλληλοι ε, προαγάγονται πολύ πιο εύκολα όταν προωθούν κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και το δικό μας μέλημα. Έχουμε λάβει πολλά παράπονα από ε, χρήστες που παραπονούνται για περιορισμό της πρόσβασης, της ανοιχτής πρόσβασης. Ακούσαμε κάτι τέτοιο και από τον κύριο Γιώχανσον. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος με πάρα πολλά επιχειρησιακά μοντέλα και δεν θα πρέπει να διευκολύνουμε ορισμένα μόνο, ειδικά τα μεγαλύτερα. Είναι σημαντικός αυτός ο πλούτος. Η πρόσβαση ε, του, του διαδικτύου ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές στη Ήπεθρο είναι πολύ θετικό. Γιατί στις χώρες που έχουμε ισχυρές τηλεπικοινωνίες ε, δυστυχώς έχουμε χαμηλή πρόσβαση. Στο Βέλγιο για παράδειγμα που για πολύ καιρό ε, φύση το προβλήματα. Μόνο το 2013 έχει εφαρμόσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να διαπιστώσει αν 400.000 ε, πολίτες μπορεί να ε, εφαρμόσουν το σύστημα στο σπίτι τους. Αυτό το κάναμε ήδη από την, από το, στην δική μου χώρα από το, από το 1990. Η καθυστέρηση του Βελγίου στον τομέα αυτό οφείλεται στο μικρό αριθμό των παρόχων υπηρεσιών και στις, στα λίγα ενάψματα που δίνονται. Να φέρω και το παράδειγμα της Ρουμανίας. Είχα πάει το 2011. Έχουν ε, εκτεταμένη πρόσβαση ακόμη και σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 75 Mbit το δευτερόλεπτο οπότε το θέμα δεν είναι κανεί μια πλούσια ή φτωχή χώρα. Το θέμα είναι τι επενδυτική πολιτική και στρατηγική ακολουθεί. Και λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ασχολείται μόνο με τις μεγάλες ε, εταιρείες. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα καινοτόμε επιχειρησιακά μοντέλα, ίσως των πιο νέων ε, χωρών μελών. Γιατί οι πιο αποτελεσματικές εταιρείες είναι οι μικρότερες που προσφέρουν και υψηλή ανταγωνιστικότητα και σχετικά χαμηλές τιμές. Οπότε φοβούμαι ότι με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά θα αναχαιτήσει την πρόοδο συγκεντρώνοντας τον έλεγχο στους λίγους και αφαιρώντας την εμπιστοσύνη από τις τοπικές αρχές που μέχρι τώρα έχουν δείξει πολύ καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη συνεργειών. Εγώ πιστεύω ότι οι τοπικές αρχές εξασφαλίζουν καλύτερη συνέργεια μεταξύ των υποδομών και Είχαμε πολύ καλά παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την τελευταία πρόταση ουσιαστικά θα υπονομευθούν οι προσπάθειες των τοπικών αρχών που στόχο έχουν την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση και σύνδεση των Ευρωπαίων πολιτών στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Έχω πάρα πολύ καλά νέα. Έχω καλά νέα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Τελκαστήγιο για να μας ενημερώσει. Ε, remind me all times. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέλφους. Και καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Χέρτσοκ για την εξαιρετική δουλειά. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα διεξοδικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και παρουσίασε και εξαιρετική δουλειά ως αποτέλεσμα. Δεν θα ήθελα να μπω τώρα τόσο πολύ σε λεπτομέρειες, αλλά να τονίσω τις δυσκολίες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Εμείς και εσείς οι σκιώδεις συζητητές όσοι ασχολούνται στενότερα με το θέμα, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει αυτή την πρόταση ως κανονισμό και αν κατάλαβα καλά υπάρχει στήριξη στις ε, τροπολογίες για οδηγία και όχι κανονισμό και ήμουν μία από εκείνους που στήριξαν ε, την οδηγία και όχι τον κανονισμό. Από την άλλη όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόταση κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την διαδικασία προσαρμογής του να γίνει ο κανονισμός οδηγία. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι πολύ δύσκολο και ορισμένες τροπολογίες υποβλήθηκαν με το σκεπτικό ότι πρόκειται για κανονισμό και όχι οδηγία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι είναι εν η διαδικασία και χρειάζονται αναθεωρήσεις κατά τη διάρκεια συζήτησης των τροπολογιών. Και να σε ευχαριστήσω ξανά, Edit, για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Εάν όχι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Υπάρχει κανείς? Εδώ είστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Βολφτίτριχ Κρούσμαν. Έχω ήδη βρεθεί στην Επιτροπή σας άλλη μια φορά. Και είμαι αρμόδιος για αυτήν την πρόταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια τη πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τι τροπολογίε, θα ήθελα να εστιάσω σε ορισμένες αρχές που διέπουν την πρότασή μας. Και να σας υπενθυμίσω τις αρχές αυτές. Καταρχάς, αναγνωρίζουμε την μεγάλη σημασία που έχει δοθεί στην πρότασή μας από αυτήν εδώ την Επιτροπή και αυτό φαίνεται με την ε, ταχύτατη εξέταση της πρότασης. Αυτό φαίνεται και από τις ε, συνεισφορές που ακούσαμε σήμερα και από τις ε, προτάσεις και φαίνεται επίσης και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο συζήτησε την πρόταση αυτή πρόσφατα και την θεώρησε ένα μέσο ενθάρρυνσης ε, της ψηφιακής κάτι που είναι και ένα από τους βασικούς πυλώνε ε, για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική πρόταση, πιστεύω, στα πλαίσια αυτά και πρέπει να τη δούμε ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια, ως μια πρόταση που θα προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να εξετάσει την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της κοινοβουλευτικής θητείας και να ολοκληρώσει τις συζητήσεις πριν τις επόμενες εκλογές. Πιστεύω πως είναι δυνατόν να συμβεί αυτό και θα συνάδει επίσης και με τους στόχους της πρότασης αυτής. Η πρόταση αυτή εξάλλου είναι ένα από αυτά τα μέτρα που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου. Όσον αφορά την ταχύτητα της ευρυζωνικής πρόσβασης που θα πρέπει να επιτευχθεί, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται απόλυτα το ε, γεγονός ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, η πρόταση αυτή θέλει να διασφαλίσει επενδύσεις έτσι ώστε να καταφέρει το ελάχιστο των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου. Και ένας από αυτούς του στόχου είναι μέχρι το 2020 να υπάρχει καθολική πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, υπάρχει ένα 50, υπάρχει μια ε, πρόταση 50% ευρυζωνικής κάλυψης υψηλής ταχύτητας. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε ως ε, ελάχιστο ποσοστό στα πλαίσια του ψηφιακού θεματολογίου. Γι' αυτό χρειάζεται να ορίσουμε το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Να σας πω ότι εάν φανούμε υπερβολικά φιλόδοξοι και θέσουμε υψηλούς στόχους, ενδεχομένως να χάσουμε αναγκαίες επενδύσεις, τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή έχουμε δεν θα μπορούν να συμμορφωθούν αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και των ε, υποδομών της. Αυτές οι υποδομές ε, συνεισφέρουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην επίτευξη των στόχων αυτών. Τώρα να σχολιάσω κάτι άλλο που νομίζω ανέφερε η κυρία Χέρτσογκ ε, για την ασφάλεια. Και να σας πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολούθησε τον κανόνα της ε, ουδετερότητας, υποβάλλοντας μια πρόταση που δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ε, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και να τονίσω ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη προσέγγιση. Τώρα, ένα σημείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το αν θα πρέπει να είναι η πρόταση αυτή κανονισμός ή οδηγία. Να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει διεξοδικά τις διάφορες ε, επιλογές που είχε, όχι μόνο με εκτίμηση επιπτώσεων, αλλά συζητήσαμε τις ε, πιθανές επιλογές και κανονισμού και οδηγίας και να σας πω ότι ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου το συντομότερο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ψηφιακή οικονομία. Και έχουμε προτείνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού, η οποία θα μπορέσει να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Μια οδηγία θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα χρειαστεί μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και θα οδηγήσει σε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Πιστεύω πως το επιχείρημα περί επικουρικότητας ε, για την ε, ρύθμιση σε τοπικό επίπεδο που αναφέρθηκε, ε, θέλω να σας πω το εξής. Εμείς ήμασταν πολύ προσεκτικοί και κατά την κατάρτιση της πρότασης αυτής προσέξαμε το επιχειρηματικό μοντέλο να μην εμποδίσει αλλά να οθήσει τις ε, επιχειρήσεις και να λάβει υπόψη τις διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της ανάπτυξης ε, είναι κάτι που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε σεβαστεί την ε, αρχή της επικουρικότητας. Φυσικά στην πρότασή μας προβλέπεται και κοινοβουλευτική εξέταση και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το Σουηδικό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει την πρότασή μας για διαφύλαξη της επικουρικότητας και όχι μόνο το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή των Περιφερειών έχει σταθεί στο πλευρό μας, έχουν διεξάγει και εκείνοι τις δικές τους αναλύσεις σε περιφερειακό επίπεδο και θεωρούν ότι ε, η πρόταση αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσει ε, για επικουρικότητα. Πιστεύω σε γενικές γραμμές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα ανοιχτή και θέλει να βοηθήσει τον νομοθέτη να βρει μία λύση, ελπίζω, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Και να τονίσω επίσης ότι η επιλογή του οργάνου ήταν εσκεμμένη και πιστεύω πως μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους που επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Αλλά πρέπει να είστε έτοιμοι και για την αντίθετη γνώμη. Γιατί φαίνεται ότι κρατούσα γνώμη στην Επιτροπή είναι κατά της δικής σας θέση. Ο κύριος Χόκμαρκ, συμπληρωματική παρατήρηση. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για τη συζήτηση ό,τι αφορά την ικανότητα και την ταχύτητα. Το θέμα δεν είναι να είμαστε όσο πιο φιλόδοξοι γίνεται. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σκέψεις ε, σε ό,τι αφορά ε, την, τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για τα 1400 Mbit. 30 Mbit το 2020, 100 Mbit για το 50% του πληθυσμού το 2020. Δεν είναι αρκετή αυτοί η στόχη της ευρυζωνίας, θα μας ξεπεράσει η πραγματικότητα. Γιατί αν ε, μείνουμε σε αυτούς τους στόχους, θα πέσουμε σε μία παγίδα. Γιατί επαιδείουμε ουσιαστικά σε αδύναμες ικανότητες και με μεγάλη διάρκεια που θα μας ε, ε, δέσουν χειροπόδαρα στο μέρο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο φιλοδοξούς στόχους. Όχι γιατί είμαστε υπέρ τη ύψη φιλοδοξία, αλλά γιατί οι παρόντε όχι δεν μα ικανοποιούν. Προτιμώ υψηλούς στόχους και μεγάλη ελαστικότητα παρά χαμηλούς στόχους και μικρή ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι τώρα κυρία Ευχαριστώ. Κρίμα που δεν χρησιμοποίησατε το χρόνο που δικαιώς να ο σκιώδης αλλά είπατε ότι μια και αναλάβατε την Προεδρία προσωρινά θέλετε να κρατήσετε μια ουδετερότητα. Κύριε Γιώχανσεν, ναι, θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες όσο περισσότερες γίνεται και θα ψηφίσουμε στις 28 Νοεμβρίου την οριστική έκθεση, οπότε μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, γιατί οι σοσιαλιστές είναι εκτός Βρυξελών σε αποστολή, οπότε θα έλεγα να συνενεθούμε την μέθε επόμενη εβδομάδα, πάντως εγώ είμαι ανοιχτή και συνεργάσιμη. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του κυρίου Χέκμαρτ, συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά όχι μόνο για την πρόταση αυτή, αλλά να την επεκτείνουμε σε όλους. Δεν έχω πιστεί ότι η οδηγία είναι ο σωστός τρόπος. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων ή οι υπουργοί είναι αρκετά υπέρ του, του ψηφιακού κόσμου και των ψηφιακών, του ψηφιακού περιβάλλοντος. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουμε υπονομεύσει το ψηφιακό θεματολόγιο γιατί ακριβώς περικόψαμε τους πόρους αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κανονισμό με την, ε, τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και αυτή είναι μια ουσιαστικά συμβαστική πρόταση. Αυτή η πρόταση είναι κάτι μεταξύ κανονισμού και οδηγίας, γιατί έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή, προσφέρει τεράστια ευελιξία με την παρούσα της μορφή στα κράτη-μέλη, αλλά δεν μας επιτρέπει να χάσουμε χρόνο με την μεταφορά, με την σωμάτωση στην ε, εσωτερική αναμετάξη και από τα κοινοβούλια. Αν, επικρίνουμε, ε, αν προκρίνουμε μάλλον την πρόταση για οδηγία πόσο αυστηρά θα τα κράτη-μέλη προς την εφαρμογή και πόσο θα ε, κινητοποιηθούν για την εφαρμογή. Γιατί η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, ξέρετε, που δεν ε, εφαρμόστηκε στη Γερμανία, οποία έκπληξη. Άρα ούτε και εδώ είναι λύση η οδηγία, γιατί θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη να διαχωρίσουν τη θέση και να μην εφαρμόσουν. Και αν θέλουμε πραγματικά οι πολίτες να ασθενιστούν ε, το, τα ψηφιακά θέματα και να εισχωρήσει τον ψηφιακό κόσμο θα πρέπει να, είμαστε, να διαλέξουμε τον κανονισμό. Και σε ό,τι αφορά τους στόχους, περιμένω τις συμβαστικές σας προτάσεις και ευχαριστώ α, την Πιλάρ που είπε ότι ε, δεν αρκεί ένα βήμα για να κάνω αυτή η μετάφαση από, την, ε, από τον κανονισμό στην οδηγία. Πάντως Είμαι βεβαία ότι στην εκστρατεία ενημέρωση θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί, όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί η τρίτη γενιά που είναι τα παιδιά μας πραγματικά ε, είναι αγανακτισμένα στο ότι δεν έχει γενικευθεί η ψηφιακή πρόσβαση. Και αν θέλουμε να προσελκύσουμε τους νεαρούς ψηφοφόρους, θα πρέπει να, του να τους πείσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την επιθυμία και την φιλοδοξία να γίνει ψηφιακή. κυρία Αντερστότερ. Πραγματικά χαίρομαι που οι, όσα απασχολούν την γενιά μας απασχολούν τα μέλη του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι και εμείς είμαστε αυτοί που ε, προωθούν, αν θέλετε, τις αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί ε, στην πράξη της Κομισιόν και την, ε, τα κείμενα τα οποία προωθούν είναι ότι τα τελευταία χρόνια προωθούν κείμενα τα οποία ευνοούν μόνο τις μεγάλες εταιρείες και ε, προωθούν ένα μοντέλο συγκεκριμένο για ε, τον ανταγωνισμό. Ε, και αυτό γίνεται μέσω ενός πολιτικού παιχνιδιού. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, διότι κανείς σε, σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ικανοποιημένος με την αλλαγή σχεδίων όταν όμως απευθύνεσαι σε κάποιον πρωθυπουργό και του λες τι πρέπει να κάνει κτλ. Ε, εφόσον δεν είναι ε, ειδικό στην τεχνολογία λέει, λέει ότι προφανώς αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν καλή κάλυψη στον τύπο. Ε, εμείς όμως σαν νέοι ανησυχούμε για τον τρόπο που αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας εξυπηρετεί, να μας υπηρετεί και κυρίως ε, όσον αφορά την, την ευρεία ζώνη. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζει αν θέλετε, την εμπιστοσύνη μας. Ανησυχώ επομένως. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η ψήφος για την έκθεση αυτή θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου και υπάρχουν πολλές συμβαστικές τροπολογίες που θα υποβληθούν. Περνάμε επομένως στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης πριν από τη συνάντηση των συντονιστών που είναι η συνέχεια για την ε, διαβούλευση για τις ε, top 10 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δώνα το λόγο στον κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίτσεστερ. Θέσεις εργασίας σε μικρέ και μεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Έχουν ιδιαίτερη σημασία. Παρατηρούμε τώρα ότι οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται από νέες επιχειρήσεις. Από 80, το 80% ε, το, επίσης ε, των Απασχολούμενο να απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Και πιστεύω ότι το ΕΠ που παράγουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται περίπου στο 50%. Υπάρχει λοιπόν ε, ένα πολιτισμικό στοιχείο, οικονομικό στοιχείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία, στον πολιτισμό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό δαπανών. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα με διάφορες κανονιστικές διατάξεις, με υπερβολική ρύθμιση, με κανονιστικό υπερθεματισμό. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ε, προκαλούν αυτές οι υπερβολικές ε, ε, ρυθμίσεις, ο υπολογισμός των απολαβών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το πρόβλημα υπολογισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς τους πολιτικούς να διατηρήσουμε υψηλά κοινωνικά πρότυπα και αυτό θα γίνει ενισχύοντα την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαλλάσσοντάς τες από το πρόσθετο διοικητικό και κανονιστικό άχθος. Υπάρχουν διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε υποβάλει σε συνεργασία με τους σκιώδεις Η προτεραιότητα ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μία από αυτές υπήρξε γενική συμφωνία ε, για μείωση, για προσπάθεια μείωσης του διοικητικού κανονιστικού φόρτου. Και μάλιστα ο, ένας πρώην υπουργός ε, στη Γερμανία, ο κ. Στόιμπερ, είπε ότι, το, η γραφειοκρατία δημιουργεί, σε, δημιουργεί απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προσθεθεί στο ΑΕΠ της χώρας. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, με το ότι η, για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος Μπαρόζο κατέφεραν να αναπτύξουν αυτόν τον ε, κανονισμό REFIT, το πρόγραμμα βελτίωσης καταλληλότητας και αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου. Φυσικά και όλα είναι θέμα κόστους και δεν μπορούμε να παρατηρούμε το κράτος από τη μία να επιθυμεί να μειώσει την γραφειοκρατία και από την άλλη να αυξάνει ε, τις ε, διάφορες εισφορές, ε, τα διάφορα τέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό οδηγεί σε επιβάρυνση και όχι σε ελάφρυνση των επιχειρήσεων αυτών. Πρέπει η νομοθεσία να γίνει πιο φιλική προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις καινοτόμες ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχουν ε, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν εξαιρετική δουλειά, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, περιβαλλοντικές ε, δράσεις, ανάπτυξη νέων συστημάτων ε, ίδρευσης φιλικών προς το περιβάλλον, για παράδειγμα. Ε, ευρεσιτεχνίες. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το top 10 των νομοθετικών ρυθμίσεων. Το όργανο που θα προκύψει θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να δίνει προτεραιότητα στις ε, μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις να τους ε, δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους ε, στους καταναλωτές και όχι να βυθίζονται και να βουλιάζουν στην γραφειοκρατία. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το τεστ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ο κανονικός υπερθεματισμός είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πιστεύουμε ότι χρειάζεται γνωμοδότηση και συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΕ και πιστεύω πως η συνεισφορά ιδιαίτερα της ε, ΕΟΚΕ θα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι εκεί μπορούμε να δούμε ε, τις ε, επιπτώσεις που έχει η υπερβολική γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου. Καταφέραμε να έχουμε μια πολύ καλή πρόταση και χάρη στις άριστες υποδομές που έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, στην βιβλιοθήκη για παράδειγμα, στο μεγάλο αρχείο στο οποίο μπορούσαμε να ανατρέξουμε. Η τεχνολογία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ανάπτυξη μελλοντικών θέσεων απασχόλησης. Για εμάς επίσης είναι σημαντικός ο πρώτερος έλεγχος, τον οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και επίσης ο εκ των υστέρων έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να αναφέρω επίσης ότι θα ήταν ε, πολύ καλό να αναπτυχθούν ορισμένα προγράμματα ε, παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα υπάρχουν στη Γερμανία το Mittelstands Monitor, τα οποία ε, αξιολογούν τις ε, επιπτώσεις που έχει το κανονιστικό πλαίσιο στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Είναι πολύ σημαντικό να αρθούν τα εμπόδια έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στις θέσεις απασχόλησης. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε με ποιον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, με ποιες πρακτικές χάνονται θέσεις απασχόλησης και τι επιπτώσεις έχει η γραφειοκρατία και οι νομοθετικές, ε, υπερβολικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε αυτές. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μια ευκαιρία στους ε, πολίτες με το να ελαφρύνουμε τους πολίτες από αυτές τις υπερβολικές ε, νομοθετικές ε, και κανονιστικές ρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ελάχιστος χρόνος μας έχει μείνει. Μέχρι τις 5.30 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, οπότε σας θέλω παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Ε, κυρία Αντρέ Περέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνική. Μικρή όπως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είπατε κι εσείς. Είναι σημαντικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κυρίως ε, η δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντική γιατί δημιουργούν και πολλές θέσεις εργασίας. Έχουμε το θέμα της απλοποίησης της διοικητικής. Μερικές φορές εφαρμόζαμε ε, περιοριστική πολιτική, ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, και γι' αυτό έχουμε πολύ χαμηλή χρηματοδότηση, πρόσβαση στη διδανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χαίρομαι πάντως για τις προτάσεις του εισηγητή, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, καλύτερες ε, ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν μιλούμε όμως ε, για την ανταγωνιστικότητα, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε σημαντικά πράγματα που είναι ιδιαίτερα προσφυλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα της υγείας, της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, θεμελιώδη δικαιώματα, το περιβάλλον. Είναι κεφαλαιόδου σημασία σε αυτά τα θέματα που δεν μπορούμε να τα θυσιάζουμε στο βωμό τη ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να είναι επικουρική και ανάλογη και να λαμβάνουμε υπόψη και τις απαιτήσει που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτες της. Είναι σημαντική αυτή η πρόταση ψηφίσματος γιατί ε, τροφοδοτεί τη συζήτηση για τις 10 ε, μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά να μην ξεχνούμε και τις ε, θεμελιώδεις μας απαιτήσει. Εμείς ως ομάδα θα συμβάλλουμε να διατηρηθεί και αυτό το μέλημα στο προσκήνιο. Ο κύριος Γιώχανσον. Τώρα θα ανοίξω το μικρόφωνο από την αρχή της ομιλίας μου. Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, συμφωνώ με πολλά από όσα είπε ο κύριος Ρούμπιχ Υπάρχει και μία διάσταση την οποία θα πρέπει να σκεφτούμε όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ε, τις σχέσεις ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και τον, τους καταναλωτές. Τι γίνεται όμως όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχάς ε, υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν περιγραφές μένα, αλλά και διάφορα κριτήρια κριτήρια που θα ε, επιτρέψουν να συγκρίνουμε τα διάφορα κριτήρια προέλευσης ανάλογα από τη χώρα. Γιατί ε, μπορεί να υπάρχουν κανόνες διαφορετικοί όσον αφορά την προέλευση, κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή προϊόντων, παραδείγματος χάρη. Κάτι άλλο ε, που θα ήθελα να δείξω είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και το ίντερνετ για να μπορούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παίξουν τον ρόλο τους. Θα μπορούσαμε να θίξουμε και να συζητήσουμε κάποια θέματα που αφορούν τους ιδιώτες καταναλωτές, αλλά πιστεύω ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ τους. Γιατί πολύ συχνά, όπως είπατε κύριε Ρουμπιχ και εσείς, αναφερόμαστε σε κάποιες νομικές υπηρεσίες που ε, προσφέρονται και στις, ε, στους, κατα, στους καταναλωτές, στους πολίτες, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τις χρειάζονται. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και το, τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Φόρντ, μπορείτε και εσείς να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Μετά από, πολλές, από μεγάλη εκστρατεία που κάναμε εμείς, ζητήσαμε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, βοηθήσουν, να, να, να, ζητήσουν κάποια νομοθεσία, κάποια ρύθμιση. Εδώ υποβάλλεται το κείμενο αυτό και πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ναι, εντάξει, προφανώς πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ε, εάν ε, νομοθετήσεις ε, για τον μικρό κάποια στιγμή θα αναγκαστείς να νομοθετήσεις για τον μεγάλο. Αλλά σίγουρα όμως θα πρέπει να προστατεύσεις αυτόν τον οποίος απασχολεί δύο-τρία άτομα σε σχέση με αυτόν ο οποίος απασχολεί πάνω από 100 άτομα. Για το top 10 νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για καθένα από αυτά, καμία από αυτές τις προτάσεις. Ε, η, ας πούμε παραδείγματο χάρη οι μικροεπιχειρήσεις ε, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκθέσεις υγειονομικές ε, για κάποιες εταιρείες ίσως αυτό είναι σημαντικό. Επίσης ε, για τον χρόνο εργασίας. Κάποιες ε, μικρές ε, επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις εξαιρέσεις και αυτό να το πούμε συγκεκριμένα. Ότι κάποιες εταιρείες δεν χρειάζεται, επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να σεβαστούν κάποιες, κάποια νομοθεσία, εφόσον συμφωνούν και οι εργαζόμενοι. Επίσης για το ΦΠΑ χρειάζεται μια ενιαία πλατφόρμα. Ε, η ενιαία αγορά δεν έχει σαν στόχο την, ταυτο, την, ε, την ε, ομοιογένεια, ένα μοντέλο για όλους. Όχι, υπάρχουν, ε, υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες και από εκεί πέρα αν κάποιο κράτος θέλει να προχωρήσει, δικό του θέμα είναι αυτό. Δεν χρειάζεται εμείς να επιβάλλουμε ομοιογενείς κανόνες σε όλους. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει, η δομάχη αυτή θα πρέπει να, να δίνεται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Δεν χρειάζεται η Κομισιό να προτείνει νομοθεσία για, όλους, για όλα τα θέματα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε οι οικονομικές επιχειρήσεις και δεν χρειάζεται να πάντοτε να κάνουμε συμβασμούς με την αριστερά. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Κούκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ με τι θα πει απλοποίηση ή απλότητα. Γιατί εμείς ως νομοθέτες δυστυχώς πολλές φορές περιπλέκουμε τα πράγματα και θεσπίζουμε περίπλοκη νομοθεσία, πολύ ε, δυσνόητες διατάξεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει όταν θεσπίζουμε μια νομοθετική διάταξη να λαμβάνουμε υπόψη και την εφαρμογή που είναι αναγκαία να γίνει αργότερα. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε ένα νομοθέτημα θα πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στο ρόλο των επιχειρηματιών που θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτές τις, τα νομοθετήματα και τις διατάξεις. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρούμπιχ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρηματοδότηση από το κόσμο για να δούμε πού βρίσκονται τα σοβαρότερα εμπόδια και πώς μπορούμε να τα καταργήσουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα σε κάθε ε, νομοθετική πρόταση που κάνουμε το πρώτο μας μέλημα θα είναι να καταργούμε τα εμπόδια που ταλανίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Και εγώ θα είμαι λακωνικός κύριε Πρόεδρε, υπακούντας τις συστάσεις σας. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία που επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο έργο τους. Όπως είπε ο κύριος Ρομπιχάν, το κατάλαβα καλά, έχει μειωθεί ήδη κατά 26% ε, ε, η γραφειοκρατία, ενώ ο στόχος μας ε, ήταν να μειωθεί κατά 20% μέχρι το 2013. Α με διορθώσει αν κάνω λάθο. Επίση, έχουμε την αναγνώριση από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ότι έχει περιοριστεί η γραφειοκρατία. Ε, αλλά δεν είναι αυτές οι πληροφορίες που έχω εγώ από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των ε, ε, συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συμφερόντων των εργαζομένων. Μερικές φορές τα παράπονα που ακούμε είναι ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατική η δομή των Βρυξελών και ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται για την περιορισμό της γραφειοκρατίας είναι αξιέπαινο και θάρεστο. Αλλά δυστυχώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θέλετε να αναγνωρίζουν ακόμη ότι έχει μειωθεί αυτό το γραφειοκρατικό άχθο. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να ζητά το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Κώστας Ανδρόπουλος, είμαι τμηματάρχης της Μονάδας για την Πολιτική ε, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της εφαρμογής ε, της ομοθετικής πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή πρόταση ψηφίσματος ε, για την οποία μπορεί να υπολογίζει στην ε, δική μας συνεργασία. Σίγουρα θέλουμε να περιορίσουμε το γραφειοκρατικό ε, άχθος και να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει αυτό εν μία νυχτή, αλλά ο στόχος είναι αξιέπαινος και τον αστερνιζόμαστε πλήρως. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιμέρους σας παρατηρήσεις σας, το πέμπτο εκτιμώντας ε, θα θέλαμε να το επικαιροποιήσουμε κάπως. Θα σας στείλουμε σχετικές παρατηρήσεις για μία ενημέρωση στο σημείο αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά το σημείο 6, σίγουρα επιδοκιμάζουμε τη, το ειδικό και υπηρεσία που έχετε για την ε, μελέτη επιπτώσεων. Θέλουμε όσο πιο στενή συνεργασία γίνεται μαζί σας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας αξιολόγηση και μελέτη επιπτώσεων, έχουμε από τον ΩΣΑ το ελεκτικό συνέδριο ε, πολύ θετικό αντίκτυπο, γιατί έχουμε από τα άργανα αυτά τις καλύτερες αξιολογήσεις ε, ε, του δημόσιου κλάδου. Πάντως ενισχύ, επικαιροποιούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της μελέτης επιπτώσεων και φροντίζουμε ώστε όλες οι ε, υπηρεσίε της, της Επιτροπής που θα προτείνουν νέες πολιτικές ε, από την αρχή θα λαμβάνουν υπόψη και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε πρόταση ενδεχομένω εκπονήσουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημείο 7, εκεί προτείνεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρεμφερές με αυτό της Γερμανίας, με τους φωτεινούς ε, σηματοδότες πράσινο, πορτοκαλί κτλ. Μα στην πράξη ήδη κάνει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί έχουμε, τις, ε, έχουμε τουλάχιστον έξι φορέ το χρόνο συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Την περασμένη εβδομάδα συναντήκαμε με έξι τέτοιε ενώσει μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκεί κάναμε μια φιλομέτρηση του προγράμματο εργασία του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014. Και εξετάσαμε ιδιαίτερα κάποιε προτάσει από το πρόγραμμα αυτό που οι μικρομεσαίε επιχειρήσει κρίνουν επαχθεί. Έχουμε δύο κατηγορίε, τι προτεραιότητε που θα τύχουν τη μέγιστη προσοχή και κατά προτεραιότητα και τις, το δεύτερο κλάδο, που θα, δεύτερο άξονα που θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ. Κύριε Ρούμπιχ, παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το 26% που αναφέρεται μείωση της γραφειοκρατίας είναι κάτι που με βρίσκει αμφίβολο. Η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση πως αυξάνεται η γραφειοκρατία και πως δεν μειώνεται. Γι' αυτό λοιπόν η ρύθμιση είναι κάτι που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε ακριβέστερα την αύξηση, την μείωση. Και μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν μέσα στις εταιρείες και ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Ευρωμαρόμετρο να ελέγξει λεπτομερώς την κατάσταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να επαληθεύσει τα ε, νούμερα που έχω στη διάθεσή μου εγώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Προθεσμία και τις τροπολογίες είναι 12 το μεσημέρι στις 7 Νοεμβρίου ή την 5η, ε, την 5η στις 12 το μεσημέρι. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρίαση αυτής εδώ της Επιτροπής και τώρα θα ήθελα να καλέσω όσους δεν θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών να καταλήψουν την αίθουσα γρήγορα και χωρίς Ευχαριστώ.